Dear colleagues, dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ να καθίσετε. Καθίστε παρακαλώ για να αρχίσουμε. Um, I, I am starting this session. Just the last warning for those. Παρακαλώ, τελευταία Ειδοποίηση για όσους ε, θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη διερμηνία. Αρχίζουμε παρακαλώ. Εξοχότητες, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, ήθιστε πια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να φιλοξενεί την εναρκτήρια σύνοδο των Open Days όπου θα συζητήσουμε το μέλλον της Ευρώπης και το πώς η πολιτική συνοχή μπορεί να βελτιώσει την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρώπη. Η Μερσέντες Πρέσο που είναι πρόεδρος Επιτροπής ε, Περιφερειών και ο Γιωχάνες Χάν που είναι αρμόδιος επίτροπος για περιφερειακή πολιτική είναι μαζί μας και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Ρόδη Κράτσα Τσακαροπούλου που είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Το Ρούντι Ντεμότ που είναι πρωθυπουργός ε, της Βαλονίας, πρόσωπος της Βελικής Προεδρίας, και τον Φιλίπ Μάιστατ, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που θα απευθύνουν ομιλίες. Επίσης ε, θα ακούσουμε και ε, μήνυμα ε, από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο. Μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσει συζήτηση με συντονιστή τον κύριο Μακ Ρότζερσον που είναι εκτελεστικός διευθυντής του Consilia Limited. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω όλους όσους ενδιαφέρονται να λάβουν το λόγο, να συμπληρώσουν τα δελτία και να τα δώσουν στους κλητήρες για να μας γνωστοποιήσουν ότι ενδιαφέρονται να μιλήσουν. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και θα ήθελα να εκφράσω την, το θαυμασμό μου για την ενεργό ανάμειξή σας στη συζήτηση για το μέλλον της ε, Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής. Νομίζω ότι ποτέ δεν είδαμε τέτοια ανάμειξη των ε, πόλεων, των δήμων, των δικτύων και των γραφείων της Οδός Βρυξέλλες και τόσο ανεκτήμητη συνεισφορά στη συζήτηση για τη μελλοντική πολιτική της συνοχής. Μάλιστα θα ήθελα να σας παρατρύνω όλους να λάβουμε την ευθύνη μας για το μέλλον της Ευρώπης γιατί εσείς προσφέρετε τον ενθουσιασμό και την ενέργειά σας που χρειάζεται η Ευρώπη και φαίνεται πρώτα απ' όλα στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και στις ευρωπαϊκές πόλεις. Σας ευχαριστώ θερμά λοιπόν που δείξατε αυτή τη μεγάλη υπευθυνότητα την αφοσίωση και δίνεται νέα πνοή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρώπη. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επομιζόμαστε και εμείς τις ευθύνες μας και προσπαθούμε να θεσπίσουμε ένα μακροοικονομικό θεσμικό πλαίσιο που θα διευκολύνει την ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων απασχόληση και την οικονομική μεγέθυνση. Είμαστε όμω πεπισμένοι ότι η Ευρώπη χρειάζεται και κάποιε διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει και μια αναπτυξιακή πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχή είναι αναπτυξιακή πολιτική και με τον κατάλληλο μακροοικονομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο μπορεί να έχει τεράστια απήχηση. Η συνοχή είναι με βάση τη συνθήκη ακρογωνίως λίθο τη ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αυτή η αρχή συνιστά την πολιτική συνοχή μια πολιτική όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Φυσικά βέβαια αυτή η πολιτική θα πρέπει να δώσει κυρίως καρπού στι περιφέρειε. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά αποτελέσματα και αυτό αποτελεί πρόκληση όχι μόνο τη πολιτική συνοχή αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για όλες τις ε, ευρωπαϊκές πολιτικές που σχεδιάζονται σε ευρωπαϊκό και εκτελούνται σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Γιατί μετά την οικονομική κρίση έχουμε νέα χαρακτηριστικά και δεν θα πρέπει να αφιστούμε προσπαθειών προκειμένου να καταλήξουμε σε μια καλύτερη και βελτιωμένη Ευρώπη. Και φυσικά θα πρέπει να γεφυρώσουμε τις ανισότητες ε, ενεργοποιώντας το δυναμικό των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών και να δώσουμε έμφαση και που χρειάζονται περισσότερες υποδομές και καλύτερες δομές. Με καλύτερη συνεργασία μπορούμε να συνδυάσουμε καλύτερα τι πιο ανεπτυγμένε περιοχέ με αυτέ που έχουν μείνει λίγο πιο πίσω. Βέβαια, όλε οι περιφέρειες και οι πόλει Ευρώπη θα πρέπει να δείξουν την ανταγωνιστικότητά τους ε, και την ισχύ τους ε, σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο. Οπότε το, ο ρόλος της εδαφικής ολοκλήρωσης είναι πολύ σημαντικό, σημαντικότερος από ποτέ. Προσθέτοντας και την εδαφική διάσταση στην ε, Ευρωπαϊκή Συνοχή, θέσαμε το δάκτυλο σε ένα ανεκτήμητο δυναμικό που μερικές φορές είναι ανεκμετάλλευτο και κρύβεται πίσω από ευρωπαϊκές και περιφερειακές στατιστικές. Το δυναμικό αυτό θα το αξιοποιήσουμε με καλύτερη προσαρμογή όλων των ευρωπαϊκών πολιτιών, ε, πολιτικών στις εδαφικές ε, ιδιαιτερότητες και στη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών και εντός της Ευρώπης αλλά και εκτός. Μια αρμονία της ευρωπαϊκής ανάπτυξης θα επιτευχθεί μόνο αν κάθε περιοχή στην Ευρώπη αξιοποιήσει το έπακρο το δυναμικό της και συνεργαστεί με τις υπόλοιπες περιοχές και εδάφη υλοποιώντας ε, τους στόχους του 2020 για, έναν, ε, μια ανάπτυξη που θα είναι βιώσιμη και ισχυρή και θα, δεν θα αποκλείει κανέναν. Είχαμε το Φόρουμ της Συνοχής από το Σεπτέμβριο του 2007 και περιμένουμε το, την 7η έκθεση συνοχής στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας υποβάλει τις ιδέες της για το μέλλον εμπνευσμένη και από τις ιδέες που θα συλλέξει στην μακρόχρονη περίοδο των διαβουλεύσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συζητήσει το ψήφισμα για το μέλλον της ε, Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής αυτή τη βδομάδα. Η μεγέθυνση και η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη θα εξαρτηθεί και από τη ζήτηση στο μέλλον. Οπότε αναπτυξιακή πολιτική και πολιτική επένδυση, ε, επενδυτική πολιτική αλλά και η πολιτική συνοχής θα έχουν ε, σημαντικό ρόλο προκειμένου να υλοποιήσουμε διαρθρωτικές αλλαγές και να πετύχουμε την ανάπτυξη για όλους. Ήθελα τώρα να προσκαλέσω την πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών, την κυρία Μερσέδες Μπρέσο, για να μας κάνει την εισαγωγική της ομιλία. Έχετε το λόγο, Μερσέδες Μπρέσο. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Χιούμπνερ, εξοχότατη, αξιότιμη κυρία Αντιπρόεδρε, κυρία Κράτσα Τσαγκαροπούλου, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Περιφερειών, Πρόεδρε Ντεμότ, Πρόεδρε Μεστάτ, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στην ενακτήρια συνεδρίαση της 8ης έκδοσης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων και στην 86η ε, Σύνοδο Λομελίας της Επιτροπής Περιφερειών. Για άλλη μια φορά η παρουσία μας και η δική μας και η δική σας σήμερα εδώ, καθώς εκείνη των 6.000 συμμετεχόντων στα 130 σεμινάρια των επομένων ημερών επιβεβαιώνουν ότι είναι σημαντικές για την Ευρώπη και οι περιφέρειες και οι πόλεις και η Ευρώπη εξίσου σημαντική για τις περιφέρειες και τις πόλεις. Σύνθημά μας είναι η Ευρώπη το 2020 ανταγωνιστικότητα, συνεργασία και συνοχή για όλες τις περιφέρειε. υπογραμμίζει αυτό αφενός την πολιτική φιλοδοξία της δικής μας σημερινής κοινή εκδήλωσης από τη μια και από την άλλη την επιθυμία να προτείνουμε στους συμμετέχοντες σε ένα βήμα ε, επικοινωνίας για θέματα που τους απασχολούν τοπικά και περιφερειακά. Το πλαίσιο, το φετινό των ανοιχτών ε, θυρών είναι σαφές. Να δώσουμε στην Ευρώπη για την επόμενη δεκαετία μια στρατηγική για το 2020 στραμμένη προς το μέλλον ε, ταυτόχρονα να φιλοδοξεί να βγάλει την Ευρώπη από την κρίση που μόλις πριν από δύο ε, ε, χρόνια άρχισε και φαίνεται θα διαρκέσει ακόμα. Δεν θέλω να είμαι υπερβολικά απεσιόδοξη, αλλά δεν μπορώ παρά να είμαι ρεαλίστρια. Δεν έχει τελειώσει η κρίση. Για να αποφύγουμε τα χειρότερα θα πρέπει να επέμβουν και τα κράτη-μέλη αλλά και οι περιφέρειες και οι τοπικές κοινωνίες. Σήμερα τα δημόσια οικονομικά υφίστανται τεράστια πίεση εργατική επισφάλεια ε, και ε, απολύσεις και οι εργαζόμενοι ζητούν τη βοήθεια του κράτους. Ε, σύμφωνα με το Δουβλίνο, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, στο δεύτερο εξάμεινο του 2010, για κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται χάνονται δύο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και απασχολεί πάρα πολύ τους Ευρωπαίους πολίτες έχουμε κάποιο περιθώριο ελιγμών, έστω και περιορισμένο. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να βλέπουμε το μέλλον ε, και το ορίζοντα του 2020, ε, έχοντας ως προτεραιότητα να βοηθήσουμε σήμερα τους ε, πιο αδύναμους. Είναι πολλές οι δυνατότητες που μπορούμε να δράξουμε και στην οικονομία της γνώσης και στην πράσινη οικονομία. Ωστόσο δεν θα πρέπει με επιπολαιότητα να δούμε τα ανησυχητικά σημεία που ακούμε από παντού γιατί ε, διακυβεύεται και απειλείται η ίδια η υγεία της δημοκρατίας μας. Δεν νομίζω ότι υπερβάλλω λέγοντας ότι η διατήρηση μιας ισχυρής συνοχής μεταξύ των περιφερειών είναι προϋπόθεση για τη συνύπαρξη στην Ευρώπη, την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ μας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Από τώρα η Ευρώπη του 2020 θα πρέπει να διαμορφώνεται με ειδικέ πολιτικές και με την απαραίτητη επαρκή χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να φτάσουμε στους φιλόδοξους στόχους που αυτή απαιτεί. Ιδιαίτερα περιμένουμε να δούμε τη νέα πράξη για την νέα αγορά, ε, την αναθεώρηση του προπολογισμού, την ατζέντα για την ευφυή απασχόληση, τις μεγάλες γραμμές της γεωργικής πολιτικής μετά το 2013 και εν τέλει την πέμπτη έκθεση συνοχής. Και άλλα σημαντικά έγγραφα που θα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους επόμενους μήνες ε, που θα αποτελέσουν μηνύματα, κατά κάποιο τρόπο θα σηματοδοτήσουν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αποτελέσουν τη βάση για τις προτάσεις για το προεπολογισμό μετά το 2013 και τα νομιθετικά ε, πακέτα του 2011. είναι στιγμή να κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί, να πούμε τι περιμένουμε εμείς από τούτη την κρίσιμη φάση. Θέλουμε να κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί, να προτείνουμε νέες ιδέες, να τις παρουσιάσουμε και κυρίως θέλουμε ε, να συμμετέχουμε ευθύς εξ αρχής. Η αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας εν μέρη οφείλεται ακριβώς και στον τρόπο που τη διαχειριστήκαμε. Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να μην ακούει, να μην αφουκράζεται τις πόλεις και τις περιφέρειές της. Η δική μας φωνή, η δική σας φωνή, συνάδελφοι, είναι εκείνη που θα ακουστεί τις ερχόμενες ημέρες στα 130 σεμινάρια, εργαστήρια, συνεδριάσεις, αλλά και με 300 δημοσιογράφους, ιδιαίτερα περιφερειακών εντύπων και μέσων ενημέρωσης που επιτέλους ήρθαν στις Βρυξέλλες και τους εύχομαι καλή επιτυχία των εργασιών για όλες τις περιφέρειες στην Ευρώπη. Ας αξιοποιήσουμε αυτή τη μοναδική ευκαιρία που έχουμε για να διατρανώσουμε τι περιμένουμε από την Ευρώπη και τι η Ευρώπη μπορεί να περιμένει από εμάς. Επ' ευκαιρία θα ήθελα εδώ να τονίσω τρία στοιχεία της συζήτησης, των συζητήσεών μας μάλλον. Πρώτον, δεν είμαστε αφελείς. Η πέμπτη ε, έκθεση για τη συνοχή και τα συμπεράσματα λέγουν ότι θα πρέπει να υπάρξει πολιτική συνοχή για όλες τις περιφέρειες όπως θέλουμε. Βεβαίως δεν μπορούμε να αναμένουμε ότι αυτό θα είναι αυτόματα ε, το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο για τον προπολογισμό. Θα πρέπει να ξέρουν από τώρα οι Υπουργοί Οικονομικοί ότι δεν ε, είναι για μας ε, εναλλακτική λύση αποδεκτή ή περικοπές στον ε, περιορισμό για τις περιφέρειες. Δεν μας ενδιαφέρουν μόνο οι λογιστικές προσεγγίσεις και οι ε, υπολογισμοί θεωρητικοί για τα διορθωτικά ταμεία. Ποιος άλλος καλύτερο από εμά ε, είναι σε θέση να ε, επιδείξει επιτυχή αποτελέσματα μετά από χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα δηλαδή αποδεικνύονται αυτά τα αποτελέσματα της πολιτικής στην πράξη. Και όπω η συνέλευση τούτη και η ίδια η Επιτροπή Περιφερειών επανειλημμένα έχουν τονίσει, η πολιτική συνοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπεται ε, να ε, είναι αντικείμενο συντονισμού μόνο σε επίπεδο κρατών μελών. Διέπεται από βασικές αρχές συγκέντρωση, ενσωμάτωση των διαφόρων τομέων πολιτικής, ε, συνεργασία μεταξύ των εταίρων και προγραμματισμός με μια κοινή στρατηγική που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης σε μια εδαφική συνοχή. Όπως Έδειξαν πρόσφατες αξιολογήσεις και αποτιμήσεις, οι αρχές αυτές είναι πιο αποτελεσματικές από ξεχωριστές τομεακές πολιτικές. Επιμέρους, η συνδίκη της Λισαβόνης δεν ορίζει τυχαία ότι ε, θα πρέπει να υπάρξει και περιφερειακή διάσταση στη συνοχή. Τρίτον, δεν είναι αρκετό οι γνώσεις και τα μηνύματα μας να παραμένουν ε, ε, γνώση και κληρονομιά κάποιων στενών κύκλων. Θα πρέπει να γίνουν γνωστά αυτά στην Ευρώπη. Αναγνωρίζω ότι έχουν γίνει πολλά τα τελευταία χρόνια για να ε, προβάλλεται καλύτερα το αποτέλεσμα της πολιτικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό την έννοια αυτή και προς το σκοπό αυτό σημαντικό στοιχείο της σημερινής συνεδρίασης ήταν ακριβώς να δείξουμε και το τοπικό στοιχείο με το σύνθημα Ευρώπη ε, στην περιφέρειά μου, η Ευρώπη στην πόλη μου που προβλέπει, και αυτό είναι μια σημαντική καινοτομία, περίπου 260 συνεδριάσεις και συναντήσεις που διοργανώνονται στις ε, περιφέρειες και τις πόλεις που είναι partner των ε, Open Days. Νομίζω ότι μπορούν ακόμα να γίνουν πολλά. Κάθε χρόνο να προχωρούμε χρησιμοποιώντας και τη σημερινή εμπειρία. Μια Ευρώπη που δεν θα είναι σημαντική για όλους και για όλα, για τους πάντες και τα πάντα, δεν θα είναι σημαντική για κανέναν. Και όπως είπε και ο Ντελόρ, ότι αν δεν προχωράς στην Ευρώπη τελικά, πέφτεις, γιατί είναι σαν ποδήλατο οι ε, περιφέρειές μας και οι πόλεις μας έχουν αρκετή ενέργεια και αρκετές ιδέες για να μπορούν να κάνουν την Ευρώπη να προχωρήσει. Ας το κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε αυτό. Είμαι ε, βέβαιη ότι η σημερινή συνεδρίαση και τις επόμενες μέρες θα έχουμε πολύ σημαντικά και πολύ ενδιαφέροντα και ελπίζω και χρήσιμα αποτελέσματα και συμπεράσματα όχι μόνο για τις περιφέρειες και τις πόλεις αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και σας ευχαριστώ που ήρθατε να εργαστείτε μαζί μας. Uh, Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μεσέντες Μπρέσο. Τώρα ο Επίτροπός μας, Γιωχάνες Χάν, υπεύθυνο για την περιφερειακή πολιτική, θα πάρει τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας ε, καλωσορίσω στην 8η έκδοση των ανοιχτών ημερών στις Βρυξέλλες. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη μεγάλη προσέλευση από τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, αρχές, ο ακαδημαϊκός κόσμος, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι επιχειρήσεις εκπροσωπούνται και θα ήθελα να σας καλωσορίσω να καλωσορίσω και εκπροσώπους χωρών όπως η Βραζιλία, η Ρωσία, η Αργεντινή, η Αρμενία, ε, που αποδίδουν μεγάλη σημασία στην περιφερειακή πολιτική και έχουν καταδείξει πόσο ε, σημαντικό είναι για αυτούς ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούμε την περιφερειακή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές, ε, δημοφιλής εκδήλωση, 130 σεμινάρια, 160 εκδηλώσεις ολόκληρη την Ευρώπη και φέτος είμαι πεπισμένος ότι θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία το εγχείρημα. Ε, η Ευρώπη 2020 και η οικονομική πολιτική, αυτό είναι το φετινό θέμα. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, πληγήκαμε από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Ε, και βλέπουμε κάποια ισχνά σημάδια ανάκαμψης. Ε, δεν μπορούμε να ε, επαναπαυθούμε. Πρέπει να ορίσουμε τις προτεραιότητές μας, να βρεθούν θέσεις εργασίας, να ανοίξει ακόμη περισσότερο η εσωτερική αγορά, δηλαδή το μεταρρυθμιστικό θεματολόγιο της Ευρώπης 2020 θα τονώσει την ανάκαμψη με τρόπο ώστε να δημιουργηθεί μια ευφιέστερη, πρασινότερη οικονομία στην οποία θα συμμετέχουν όλοι. Ε, οι περιφέρειε και οι πόλεις ε, θα διαδραματίσουν καταλητικό ρόλο και αυτό εξ αρχή. Είναι φιλόδοξη η στόχη μας ευρωπαϊκό επίπεδο για την Ευρώπη 2020 με επενδύσει 3% του ΑΕΠ ε, για την έρευνα και την ανάπτυξη. Έχουμε τους κλιματικούς στόχου. επίσης τους στόχου για την απασχόληση, την παιδεία, την μείωση της φτώχεια. Όλοι αυτοί οι στόχοι πρέπει να μετατραπούν σε περιφερειακού στόχου. Κάθε περιοχή θα έχει διαφορετικό στόχο, γιατί έχει διαφορετικό δυναμικό, διαφορετικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει για να εκπληρώσουμε τι κοινέ φιλοδοξίε μα. Βασικοί φορεί από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα θα συμμετάσχουν, ώστε αυτέ οι φιλοδοξίε να μεταφραστούν σε πρακτικά μέτρα. Οι ανοιχτέ ημέρε είναι ιδανική πλατφόρμα προβληματισμού για να διαμορφώσουμε από κοινού το μέλλον μα, για να συνεργαστεί καλύτερα ιδιαίτερα ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας, οι επιχειρήσεις δηλαδή, ούτως ώστε να κάνουμε τη διαφορά. Γνωρίζετε ότι τον επόμενο μήνα θα υποβάλουμε την πέμπτη έκθεση συνοχής. Ε, θα δούμε λοιπόν το πανόραμα της μελλοντική πολιτικής συνοχής και με τις προτάσεις μας θέλουμε να αρχίσει η ευρεία διαδικασία διαβούλευση και τον Ιανουάριο θα διοργανωθεί το αντίστοιχο φόρμου, ώστε να δούμε πώς ε, με συνεχή τρόπο θα μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στις ραγδαίες εξελίξεις ε, του οικονομικού τοπίου. Σήμερα θα ακούσουμε τη φωνή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όλων των περιφερειών ε, για να ακούσουμε, να εισακουστούν οι επιθυμίες σας για το μέλλον. Ε, ευχαριστούμε την Επιτροπή των Περιφερειών, τον βασικό έταρο για τη συνεχή συμβολή του. Το ίδιο ισχύει και για του συναδέλφου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που με τι εκθέσει του συνέβαλαν τα μάλα στην διαμόρφωση τη μελλοντική πολιτική και στον προβληματισμό μας. Ευχαριστώ και τη Βελική Προεδρία για τον επαγγελματισμό τη και την αφοσίωσή τη, διότι προώθησε αυτή την πολιτική και υπολογίζουμε στη βοήθειά σα ούτω ώστε τα παροσυχία να μπορέσουμε να εγκρίνουμε του απαιτούμενου κανονισμού. Επίση, Επίσης, ε, είναι θέμα συνεργασίας, ε, δηλαδή έχουμε τοπικές ιδιομορφίες, ε, αλλά με, μια, με έναν ευφυή συντονισμό των πολιτικών και των μέτρων μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Εγώ μετέβη σε διάφορες περιφέρειες και εξεπλάγει από τις καινοτόμες ιδέες και από το ευρύ φάσμα προγραμμάτων που υποστηρίζονται από την Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επόμενες ημέρες θα παρουσιαστούν πολλά από αυτά τα σχέδια και θα δράξουν κοιτάξουμε αυτή την ευκαιρία για να μάθουμε από τους άλλους, να εμπνευστούμε. Σας εύχομαι να είναι υπέροχες οι επόμενες ημέρες εδώ στις Βρυξέλλες. Thank you. Thank you, Ευχαριστούμε, Επίτροπε Χάν. Τώρα η κυρία Κράτσα Τσαγαροπούλου, ε, η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρακαλείται να προσέλθει στο βήμα για να κάνει την αγόρευσή της. Κύριε Επίτροπε, αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική, αγαπητέ κύριε Χάν, Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Περιφερειών, αγαπητή κύριε Μπρέσο, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αγαπητέ κύριε Μέιστατ, κύριε Πρωθυπουργέ της Βαλονίας, αγαπητέ κύριε Ντεμότ, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρώην Επίτροπε Αρμόδια για θέματα Ευρω... περιφερειακής πολιτικής. Κυρία Χιούμπνερ, αγαπητοί συνάδελφε, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα ως Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να εκπροσωπήσω το θεσμικό μας όργανο και τον πρόεδρο του, τον κύριο Γέζη Μπούζεκ, σε αυτή την 8η εβδομάδα των περιφερειών και πόλεων, τις ανοιχτές μέρες για το 2010. Αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2003 και αποτέλεσε συνδιοργάνωση της Επιτροπής Περιφερειών και της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με 244 περιφέρειες και πόλεις από 33 διαφορετικές χώρες. Η συνεργασία αυτή έχει έναν εκτίμητο πλεονέκτημα. Μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε από κοινού και σε υψηλό επίπεδο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής. Επίσης μας επιτρέπει η συνεργασία αυτή να αξιοποιήσουμε καλύτερα τον πλούτο, τις δυνατότητες και το δυναμικό των ευρωπαϊκών περιφερειών και πόλεων. Η πολιτική συνοχή, αγαπητοί φίλοι, αποτελεί έναν σημαντικότατο στόχο της ευρωπαϊκής ε, πολιτικής και του ευρωπαϊκού οράματος γιατί με ορατό και απτό τρόπο καθώς και με πόσο τικοποιημένο τρόπο απηχεί την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Ο στόχος της πολιτικής συνοχής ήταν ανέκαθε να συμβάλλει στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη των κρατών μελών και των περιφερειών, ιδιαίτερα των λιγότερων ανεπτυγμένων, προσανατολισμένη προς την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα όλων των περιοχών, προσπαθώντας να προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Μετά από τις διαδοχικές διευρύνσεις της ε, Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτική συνοχής χρειάστηκε να εγκληματιστεί και να προσαρμοστεί διαδοχικά σε διάφορες πραγματικότητες και σε πολύ σημαντικές ε, περιφερειακές διαφορές όπως υπεραπόμακρες περιοχές ή ιδιαίτερα βιομηχανικές περιοχές ή αεροκατοικημένες περιοχές, οι νησιωτικές περιοχές και περιφέρειες. Η περιφερειακή πολιτική προσπαθεί να φέρει την Ευρώπη κοντά στους πολίτες και προσκαλεί τους εταίρους της σε διάφορα επίπεδα να συνεργαστούν. Μάλιστα η πολιτική αυτή είναι ορατή και προσιτή ε, προς τους πάντες και αποτελεί μία από τις ε, πλέον προσφυλείς πολιτικές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέβαλε τα μάλα στην διαμόρφωση της πολιτικής συνοχής της περίοδου 2007-2013. Και μάλιστα ενισχύοντας πρώτα απ' όλα την ε, διακρατική και τη διαπεριφερειακή συνεργασία και δίνοντας έμφαση στη χρήση των κονδυλίων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε μια αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος χωρίς ταυτόχρονα να μελεί την προώθηση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας, της ισότητας των ευκαιριών και της κοινωνικής ένταξης. Πρόσφατα αντιμετωπίσαμε νέες προκλήσεις ε, στην οικονομική μας ζωή και χρειάστηκε να λάβουμε με νέα μέτρα προκειμένου να επιταχύνουμε την εφαρμογή των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007 και 2013. Προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε όλους τους πόρους και τα μέσα προκειμένου με αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο να στηρίξουμε τις προσπάθειες ανάκαμψης που γίνονται σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Και από την άποψη αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταρτήσει μια έκθεση και έχει γκρίνει ένα ψήφισμα που αφορά την συμβολή της περιφερειακής πολιτικής της Ένωσης στην καταπολέμηση της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης, ιδιαίτερα στα πλαίσια του στόχου 2. Και μάλιστα ε, επί τη ευκαιρία αυτή είχα τη δυνατότητα ως μέλος της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως εισηγήτρια για το θέμα αυτό συνέβαλα και εγώ στην ε, ανάληψη αυτής της πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας. Οι ανοιχτέ ημέρες του 2010 ε, προσανατολίζονται την Ευρώπη του 2020, την ανταγωνιστικότητα, τη συνεργασία και τη συνοχή για όλες τις περιφέρειες. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2020 προσβλέπει σε μία έξυπνη, αηφόρο, φιλόδοξη και αλληλέγγυα ανάπτυξη. Φυσικά κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την επιτυχία της στρατηγικής του 2020 και μια επιτυχημένη πολιτική συνοχής. Όπως είπε και ο ο Μάριο Μότη στην υποβολή της εκθεσής του για την στρατηγική του 2020. Η στρατηγική αυτή επιβεβαιώνει ότι η πολιτική συνοχής ε, είναι σημαντικό στοιχείο και προτεραιότητα, προτεραιότητα όλων των ευρωπαϊκών πολιτικών και τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν κέριο μηχανισμό για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς συμπεριλαμβανομένου του στόχου και της κοινωνικής ένταξης. Η περιφερειακή διάσταση λοιπόν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και στην πρόταση για την αναθεώρηση του κοινοτικού προϋπολογισμού και τη διαμόρφωση του μελλοντικού δημοσιονομικού πλαισίου. Μία ισχυρή και επαρκώς εφοδιασμένη με οικονομικά μέσα περιφερειακή πολιτική αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να υλοποιήσουμε το στόχο της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Μάλιστα, μία, α, ένας καλύτερος συντονισμός και συμπληρωματικότητα με τους εθνικούς προϋπολογισμούς είναι απαραίτητες προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τα αποτελέσματά μας. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε και τη σημασία που έχει εδώ η ελαστικότητα προκειμένου να προσαρμόσουμε τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες και τη στήριξη στις επιμέρους περιφέρειες στις οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Και αυτό ισχύει και για τις ε, υπεραπόμακρες περιοχές, για τις παραμεθόριες περιοχές ή τις περιφέρειες που έχουν ε, ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπως είναι οι νησιωτικές ε, περιφέρειες και οι ορεινές περιοχές. Μάλιστα, μια προσέγγιση που θα καλύπτει και τη διάσταση των πόλεων σε την πολιτική συνοχή είναι απαραίτητη. Γιατί και οι πόλεις διαδραματίζουν σήμερα έναν πολύ σημαντικό και δυναμικό ρόλο στην ανάπτυξη των περιφερειών και δίνουν μια όθηση, θετική όθηση στην ε, οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Οπότε η πραγματικότητα είναι πολυεπίπεδη και πολυσύνθετη. Ως εκ τούτου είναι επιτακτική ανάγκη την επόμενη περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού να προβλέψουμε τους απαραίτητους πόρους για τις επενδύσεις στα διάφορα προγράμματα για τις πόλεις και θα πρέπει και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πόλεις να είναι συνεπής, συνεκτική και να περιλαμβάνει όλες τις πόλεις. Θα πρέπει έτσι να προσθέσουμε μια σημαντική προστιθεμένη αξία και η πολιτική μας να εφαρμόζεται χάρη στην ε, τοπική στήριξη αλλά και στις ε, γνώσεις και το δυναμικό των περιφερειών. Θα πρέπει να δώσουμε μια συντονισμένη απάντηση από πλευράς και των περιφερειών και των κρατών μελών. Και εκδηλώσεις σαν τη σημερινή και παρόμοιες διοργανώσεις με συμμετοχή πολιτικών ηθινόντων, εκπροσώπων των τοπικών και περιφερειακών αρχών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, εμπειρογνωμόνων ε, και ακαδημαϊκών από όλες τις περιοχές της Ευρώπης. Η παρουσία όλων αυτών έχει κέρια σημασία σε τέτοιες εκδηλώσεις και επιτρέπει μια καλύτερη ανταλλαγή απόψεων και βέλτιση των πρακτικών προκειμένου να προωθήσουμε τις πολιτικές μας και την αγαστή συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών. Θα ήθελα κατά κλείδι να σας ε, παρουσιάσω τους στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ε, πολιτική συνοχή μετά το 2013. Η νέα πολιτική θα πρέπει να προβλέπει και ένα μεταβατικό καθεστώς που θα λαμβάνει υπόψη τις προηγούμενες εμπειρίες και τις ε, τελευταίες τάσεις και χαρακτηριστικά της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης των διαφόρων περιφερειών. Χρειαζόμαστε μια καλύτερη νομοθεσία αλλά και μια πλούστευση των κανόνων που διέπουν τα διαρθρωτικά ταμεία, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και πιο απτά αποτελέσματα και καλύτερες επιδόσεις. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, οι δικές σας ιδέες και προτάσεις Όλες οι συνεισφορές που θα συγκεντρώσουμε σε αυτές τις ανοιχτές μέρες θα είναι πολύτιμες για να, βελτιώσουμε και να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά μια περιφερειακή πολιτική και πολιτική συνοχή. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμβολή σας, την προσοχή σας, την αφοσίωσή σας και σας εύχομαι καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Αντιπρόεδρε. Επόμενος ομιλητής είναι ο Πρωθυπουργός Περιφέρειας της Βαλονίας, κύριος Ρουντί Ντεμότ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Περιφερειών, κύριε Επίτροπε Περιφερειακής Πολιτικής, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής του Κοινοβουλίου, κύριε Μεστάτ, Κυρίες και κύριοι, είναι για μένα μεγάλη τιμή ευκαιρία που έχω να εκπροσωπώ τη Βελγική Προεδρία στα πλαίσια της έναρξης της 8ης ε, ε, εκδοχής των ε, ανοιχτών ημερών. Πρώτον, γιατί από μόνη της η εκδήλωση αυτή έχει νόημα, κινητοποιεί και είναι και καρπός συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Περιφερειών της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής 245 πόλεων και περιφερειών από 34 χώρες του τραπεζικού τομέα των επιχειρηματιών και της κοινωνίας βεβαίως των πολιτών. Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι στα 8 αυτά ε, χρόνια ε, ε, οι μερίδες που διοργανώνονται, οι ανοιχτές ημερίδες ε, έχουν δοκιμαστεί και αποδειχθεί ε, στην πράξη αποτελεσματικές. Οι πόλεις και οι περιφέρειες έδειξαν το ενδιαφέρον τους και διαδραματίζουν και πρωταγωνιστικό ρόλο ε, προωθώντας τον επικοδομητικό όσο και διαρκή διάλογο των Ευρωπαίων πολιτών με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ευαισθητοποιούν το κοινό και ενημερώνουν περισσότερο για τις προκλήσεις που άμεσα το αφορούν. Και τέλος, ενισχύουν και αναπτύσσουν συνεργασίες με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Για μένα όμως είναι και χαρά ευκαιρία που έχω να συμμετέχω εδώ ε, ενώπιον σας σήμερα. Γιατί η άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου είναι θαυμάσια ευκαιρία και προνόμιο για μια χώρα. Πόσο μάλλον μια χώρα ομοσπονδιακή όπως είναι το Βέλγιο. Δίδεται η ευκαιρία, η μοναδική ευκαιρία να συμμετέχουν ε, τα ομόσπονδα ε, κράτη σε αυτή την προσπάθεια και να δείχνουν την εμπειρία τους και την τεχνογνωσία τους. Είναι επίσης και μια ευκαιρία για τους εταίρους για να θυμίσουμε ότι ο βαθμός της ευβάθυνσης ε, του βελγικού φεντεραλισμού δίνει στις περιφέρειες ε, στο Βέλγιο όχι μόνο μεγάλη αυτονομία και αυτοτέλεια αλλά και τη νομική υπόσταση για διεθνή παρουσία. Τέλος, είναι μεγάλη τιμή η ευκαιρία που έχω εδώ να παρευρίσκομαι ενώπιόν σας αν σκεφτώ τα θέματα που επιλέξατε. Ανταγωνιστικότητα, συνεργασία αλλά και συνοχή. Πρέπει να σας πω ότι η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μεγάλη προτεραιότητα της Βελγικής Προεδρίας. Γνωρίζετε ότι η Προεδρία δεν εκφέρει γνώμη, δεν συμμετέχει στις συζητήσεις βεβαίως, αλλά ε, χαράσει προτεραιότητες και το μέλλον της πολιτικής συνοχής για την περίοδο μετά το 2013 συνιστά προτεραιότητα. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια περίοδο μεταρρυθμίσεων, μετάβασης και μετασχηματισμού. Από τη μια χρειάστηκε να διανύσει κρίση που βεβαίως έχει επιπτώσεις ως προς την ανεργία, τις κοινωνικές ανισότητες, αλλά ταυτόχρονα η κρίση αυτή κατέδειξε διαρθρωτικές αδυναμίες της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αφετέρου, αυτή η περίοδος μετασχηματισμού απορρέει από την απάντηση που πρέπει να δώσουμε στην παγκοσμιοποίηση, στην πίεση των φυσικών πόρων και στη δημογραφική πίεση και εξέλιξη. Υπό την έννοια αυτή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθύμησε ότι ο στόχος κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής παραμένει περισσότερο από ποτέ στο κέντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η ε, πολιτική συνοχής είναι μοχλός, για να μην πω πρωταγωνιστής, για να επανέλθει η διαρκής βιώσιμη ε, αηφόρος και ισόρροπη ανάπτυξη αλλά στο σύνολο της ευρωπαϊκής επικράτειας. Τα διαρθρωτικά ταμεία είναι βασικός και ισχυρός φορέας συνοχής για τις περιφέρειες και τις πόλεις στην Ευρώπη. Η παρέμβαση των ταμείων αυτών ε, επιτρέπει μακροχρόνια και δημιουργία θέσεων απασχόλησης αλλά και ωφέλη για τις περιφέρειες. Επίσης τα διορθωτικά ταμεία μπορούν να είναι ένα βασικό εργαλείο εφαρμογής της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020. Είναι λοιπόν άκρος επιθυμητό αυτή η δυνατότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα να δρά μέσω των διαστατικών ταμείων όχι μόνο να διατηρηθεί αλλά και να ενισχυθεί. Είναι εκ των όνου κάνευια τη συνέχιση μιας ισόρροπης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. από τις βασικότατες προτεραιότητες και της Βελγικής Προεδρίας ε, του Συμβουλίου της Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, Πρόεδροι, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι η ε, σημερινή συζήτηση γίνεται σε μια συμβολική συγκυρία. Γιατί για το μέλλον της πολιτικής συνοχής παίζει κρίσιμο ρόλο. Λίγες είναι εβδομάδες που μας χωρίζουν από την έγκριση του, της πέμπτης έκθεσης για τη συνοχή που θα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση αυτή θα δώσει μια εμπεριστατωμένη ανάλυση της κατάστασης και θα βάλει και κάποια ορόσημα, για παράδειγμα, που βρισκόμαστε, μια αποτίμηση ως προς τη σύγκληση των οικονομιών. Να γνωρίζουμε πώς συνεισφέρει και συμβάλλει η πολιτική αυτή στους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς διαρθρώνεται και διασυνδέεται και με τις άλλες πολιτικές, και τις ευρωπαϊκές και των κρατών μελών. Και θα περιέχει η έκθεση αυτή και κάποιους πρώτους προσανατολισμούς για το τι ε, μοίρα θα επιφυλαχθεί στην πολιτική συνοχή μετά το 2013. Αμέσως μετά την πέμπτη έκθεση η Βελγική Προεδρία θα ε, διοργανώσει άτυπο ε, συμβούλιο των Υπουργών που ασχολούνται με αυτά τα θέματα στη Λιέγη 22-23 Νοεμβρίου. Θυμίζω ότι απευθύνθη στην Επιτροπή Περιφερειών ως Βελγική Προεδρία για τη σύνδεση της ε, διαρθρωτικής πολιτικής με τη στρατηγική του 2020. Πάρα πολύ σημαντικό. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να χαράξουμε την ε, μελλοντική πολιτική για καλύτερη ισορροπία της συνοχής και θεματική και εδαφική. Μέσω αυτών των θεμάτων θα πρέπει να αναλύσουμε ε, τις απαντήσεις που δίνουμε στην πολιτική συνοχής και ε, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που σήμερα ε, έχει να ε, ξεπεράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό, εδαφικό αλλά ξέρουμε ότι είναι περιορισμένες οι προτεραιότητες ε, κάθε φορά και θα, πρέπει επαναλαμβάνω να δούμε πώς συνδέεται η πολιτική συνοχή με, με άλλες κοινοτικέ πολιτικές με τη στρατηγική το 2020 και να δούμε ποιες προτεραιότητες θα χρειαστούμε ε, και στην πολιτική συνοχή υποστήριξη της καινοτομία και της οικονομίας της γνώσης. Τα ίδια ισχύουν και για την απασχόληση και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ε, ικανοτήτων που είναι και στοιχεία κοινωνικής συνοχής πώ μπορεί να συμμετέχει η συνοχή για την αηφόρο βιώσιμη ανάπτυξη, για τη στρατηγική 2020, για μια πιο πράσινη οικονομία, πιο ανταγωνιστική, με πιο ορθολογική χρήση των φυσικών μας πόρων. Κυρίες και κύριοι ε, πρόεδροι, Κύριε Επίτροπε, τελειώνοντα, ήθελα να ευστήσω την προσοχή στην προτεραιότητα που δίνει η Βελγική Προεδρία ε, στη συνοχή η προηγούμενη προγραμματική περίοδος των διαστατικων ταμειων ταμείων 2007-2013 ε, βασίστηκε στη συνοχή, την ενίσχυσε και ε, προέβλεψε ένα εργαλείο που έχει σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και θα πρέπει να διατηρηθεί. Ας θυμίσουμε τι έγινε. Τα ευρωπαϊκά δίκτυα, η ανάπτυξη συνεργασία, ε, ε, η καινοτομία και η εμπειρία στα διάφορα επιμελητήρια. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια της συνοχής και της συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών. Αυτό ακριβώς απασχόλησε μια υψηλού επίπεδου διάσκεψη που διοργάνωσε η Βελγική Προεδρία στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 ε, Οκτωβρίου στο Τουρνέ. Η ε, ε, διάσκεψη αυτή του τουρνέ ήταν από μόνο του ένα αποκεντρωμένο γεγονός και μια εκδήλωση των Open Days. Ευχαριστώ την κυρία ε, Μπρέσο, την κυρία Χιούμπνερ, τον Επίτροπο κύριο Χάν για τη συμμετοχή τους και μάλιστα την ενεργή συμμετοχή τους. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης αυτής εξεταστήκαν ιδιαίτερα θέματα όπως είναι η σύνδεση μεταξύ της εδαφικής συνεργασίας και της στρατηγικής 2020. Η, η, και αναθεώρηση του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία με συγκεκριμένες προτάσεις και θα ήθελα να σας επισημάνω ότι αν επιθυμείτε υπάρχουν και οι εκθέσεις ζητήστε από τη γραμματεία. Να σας ενδιαφέρει. Κυρίες και κύριοι, η συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραματίζουν στην Ευρώπη οι περιφερειακές και τοπικές αρχές. Η ευρεία ε, επέκταση της αρχής επικουρικότητας και οι μηχανισμοί που προβλέπονται επιτρέπουν ε, στις αρχές αυτές να ε, ελέγχουν και την καλή υλοποίηση των πολιτικών αυτών. Είμαι απολύτως στη διάθεσή σας και ε, πιστεύω στη σημαντική αποστολή που έχουμε να διατηρούμε διάλογο μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Και μπορείτε να υπολογίζετε στη Βελγική ε, Προεδρία που βλέπει το ρόλο της ως διαμεσολαβητή, ως διευκολυντή του διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστούμε. Τώρα θα ήθελα να ζητήσω από τον Επίτροπο χάνο μας παρουσιάσει το μήνυμα μέσω βιντεοδιάσκεψης που μας στέλνει ο Πρόεδρος Μπαρόσο. Ο πρόεδρος ε, Μπαρόσο μου είπε να σας δηλώσω πόσο λυπάται που δεν μπορεί να έρθει σήμερα ε, φυσικά αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο των περιφερειών, ειδικά σε αυτή την περίοδο και γι' αυτό επέμεινε για να μας στείλει ένα βίντεο μήνυμα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, ήθελα πραγματικά να συμμετάσχω στις ανοιχτές ημέρες του 2010, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Ε, δυστυχώς όμως κολλείομαι σήμερα και λυπούμε ειλικρινά. Γι' αυτό το λόγο επέμεινα να σας στείλω αυτό το μήνυμα. Η Ευρώπη εδώ και δύο χρόνια υφίσταται σοβαρή πίεση λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Παρόλα αυτά, ε, καταλήξαμε σε κάποιες λύσεις, μπορέσαμε να χτυπήσουμε τα προβλήματα στη ρίζα τους, ενισχύοντας την οικονομική διακυβέρνηση και συντονίζοντας τις οικονομικές πολιτικές μας, καθώς και μέσω ε, χρηματοπιστωτικών ρυθμίσεων. Από κοινού έχουμε καταφέρει πάρα πολλά και τώρα ε, βαδίσουμε σε πιο σταθερό έδαφος. Έχουμε καλύτερες οικονομικές προοπτικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ξεκινήσει η ανάκαμψη και παρότι παραμένει σε υψηλά επίπεδα η ανεργία, ενέργεια έχει σταματήσει η αύξησή της ε, και είμαστε σε καλύτερη θέση αναμφισβήτητα σε σχέση με πριν από δύο χρόνια. Τώρα θα πρέπει να επισπεύσουμε τις προσπάθειές μας για να έχουμε αποτελέσματα μέσα από την πολιτική Ευρώπη 2020 και τις σχετικές πρωτοβουλίες. Ο στόχο μα είναι η κοινωνική οικονομία της αγορά Ευρωπαϊκή Ένωση να επανέλθει σε θετική τροχιά, ούτω ώστε να έχουμε μια ευφυή, βιώσιμη και αλληλέγγυη ανάπτυξη. Οι περιφέρειε και οι πόλεις τη Ευρώπη θα είναι βασικοί παίκτε στη στρατηγική Ευρώπη 2020. Θα παίξουν καταλητικό ρόλο, θα δημιουργήσουν νέε βιώσιμε θέσεις απασχόλησης, θα επενδύσουν σε τεχνολογίε, θα καταπολεμήσουν τι κλιματικέ αλλαγέ, θα μα δώσουν ποιοτική εκπαίδευση θα προαγάγουν την κοινωνική ένταξη, θα αναπτύξουν τις υποδομές και θα ανοίξουν το δρόμο για ευφυή ε, χωροταξική και αστική ανάπτυξη. Οι προτεραιότητες στρατηγικής Ευρώπη 2020 ε, θα έχουν κεντρικό ρόλο και στα πλαίσια δύο βασικών πολιτικών οροσίμων που σας αφορούν άμεσα. Πρώτον, η ανθεώρηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σύντομα θα παρουσιάσει τις αρχικές της σκέψεις επ' αυτού. Δεύτερον, η συζήτηση για την πολιτική συνοχή μετά το 2020 2013 που θα λάβει η χώρα τους προσεχείς μήνες. Αυτά τα δύο βασικά ζητήματα θα είναι μια πραγματική δοκιμασία για μας. Πρέπει να περιμνήσουμε ούτω ώστε να γίνονται με πιο αποτελεσματικό τρόπο οι δαπάνες μας, να αυξήσουμε την, προσ... την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να απλουστεύσουμε την εφαρμογή των νομοθετημάτων. Φυσικά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη δημοσιοοικονομική πίεση, αλλά θα ήθελα να ξεκαθαρίσω το εξή. Οι βασικέ αρχέ τη πολιτική συνοχή θα παραμείνουν αναλύωτε. Αυτή η πολιτική είναι η έκφραση Τη της ευρωπαϊκής πολυλεγγύης ε, που βρίσκεται στον πυρήνα της διαδικασίας ολοκλήρωσης πολιτικής συνοχής ε, θα εξακολουθήσει να είναι μια στρατηγική πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και από κοινού θα αναζητήσουμε συνέργειες ε, ούτως ώστε να στεφθεί με επιτυχία η στρατηγική Ευρώπη 2020. Ε, θα ήθελα να ζητήσω την υποστήριξή σας. Είναι πραγματικά κέρια σημασία ε, να έχουμε την αμέριστη υποστήριξη των περιφερειών και των πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναπτυξιακή μας πολιτική. Ό,τι και αν μπορείτε να κάνετε. Στα κράτη-μέλη μα την τοπική κοινωνία σας για να συζητηθεί το θέμα της αλληλεγγύας, για να τονιστεί η σημασία του να έχουμε ακόμη φιλοδοξίες για τον επόμενο προϋπολογισμό της πολιτικής συνοχής της Ένωσης και για όλους αυτούς τους λόγους εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει ε, να ενισχυθεί ο διάλογος ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες. Νομίζω θα έχετε μια καλή ανταλλαγή εμπειριών ε, και γνώσεων κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών ε, και αναμένω με ανυπομονησία την έκβαση των συζητήσεών σας. Ε, ελπίζω να υποφεληθείτε από τις ανοιχτές μέρες του 2010. Yeah, Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε στην καμπή της, ε, του προβληματισμού για τη μελλοντική πολιτική, οπότε θα ήθελα να ε, απηχήσω την ομιλία του κυρίου Μπαρόζο και να σχολιάσω αυτά που είπε για τον προϋπολογισμό και για την πολιτική συνοχής μετά το 2013. Είπε ότι θα είναι μια δοκιμασία για μας. Ε, προσυπογράφω πλήρως αυτό το μήνυμα. Γνωρίζουμε όλοι πόσο σημαντική υπήρξε η πολιτική συνοχή για την περιφερειακή ανάπτυξη δεν μοιράζουμε λεφτά. Επενδυτική πολιτική καταρτίζουμε ε, και είναι κέρια η σημασία αυτή τη πολιτική, ούτω ώστε να έχουμε μια ε, ευφυή και βιώσιμη ανάπτυξη όπου θα συμμετάσχουν όλοι. 230 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν κατανεμηθεί σε βασικούς τομείς σε βάση της Ευρώπης σε 2020. Ε, έχουν τελεσφορήσει ήδη πάρα πολλές επενδύσεις σε προηγμένες τεχνολογίες, υψηλό έντερνετ ε, κατάρτιση, ευφύς, ε, τεχνολογίες, πράσινες τεχνολογίες, αλλά θα πρέπει να διατηρήσουμε τον ίδιο ρυθμό. Να έχουμε επίγνωση του ότι η πολιτική συνοχή δεν έχει μόνο υποστηρικτές, κάποιοι επιχειρηματολογούν και ισχυρίζονται ε, ότι δεν συνδέεται στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση η περιφερειακή πολιτική, ότι γίνεται άνισος καταμερισμός ε, των κονδυλίων. Ε, θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτό τον ισχυρισμό και να καταβάλουμε προσπάθειες για να βελτιωθεί η πολιτική. Η έκθεση αξιολόγησης που δημοσιεύθηκε φέτος το τονίζει αυτό. Παραμένουν μεγάλες οι και ελπίζουμε η μελλοντική πολιτική να δώσει ικανοποιητική απάντηση και σε όλα αυτά τα προβλήματα και θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε τρεις άξονες. Ε, συγκέντρωση, αποτελέσματα και ρεσιμότητα. Για την συγκέντρωση, ο πρόεδρος Μπαρόσο ήδη τόνισε πόσο ζωτικός είναι ο ρόλος της πολιτικής συνοχής, ούτως ώστε να εκπληρώσουμε τους φιλόδοξους στόχους Ευρώπης 2020. Θα ήθελα μόνο να προσθέσω ότι ε, η Ευρώπη 2020 δεν, αντικρού, δεν αντιβαίνει στην πολιτική συνοχή. Οι στόχοι της Ευρώπης 2020 ισχύουν για όλες τις περιοχές και φυσικά για, το, για τη μελλοντική επιτυχία της Ευρώπης 2020. Δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής, είναι οικονομικό το ζήτημα. Δεύτερον, μετά από τρεις γενναίες προγραμμάτων θα πρέπει να είμαστε σε θέση να ε, εξηγήσουμε με καλύτερο τρόπο στους βασικούς παίκτες ε, για ποιο λόγο δαπανούμε κονδύλια στα πλαίσια της περιφερειακής περιφερειακής πολιτικής. Γι' αυτό θα πρέπει οι περιφέρειες να ε, έχουν στόχους ε, εξακριβώσιμους, μετρήσιμους, για να μπορούμε να συζητούμε για την πρόοδο ή για την έλλειψη της πρόοδου. Είναι θέμα ευθύνης, ε, διαφάνειας, για να είμαστε όλοι υπόλογοι και έχουμε κοινά ωφέλη αλλά και κοινέ ευθύνε. Τέλος, ε, ε, με τις ε, παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις φάνηκε ξεκάθαρα ότι υπάρχουν ανησυχίες για τη σταθερότητα, για τις δομικές μεταρρυθμίσεις και για την ανταγωνιστικότητα. Είναι πραγματικά αλληλένδετες οι οικονομίες μας και εποφελούμεθα από την πρόοδο σε άλλα κράτη-μέλη, αλλά ταυτόχρονα μας πλήγουν και οι αποτυχίες τους. Ε, και γι' αυτό έχουμε αυτό το θέμα των κοινοτικών κονδυλίων ε, που πρέπει όμως να είναι συνάρτηση ε, τριών ώρων που είναι απαραίτητη για να είναι αποτελεσματικές οι επενδύσεις. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν και άλλα σημαντικά ζητήματα που πρέπει να πάρουμε υπόψη όπως ακούστηκε ήδη σήμερα, πώς να είναι απλούστερες, πιο αποτελεσματικέ οι διαδικασίες μας, πώς να μεριμνήσουμε ούτως ώστε η πολιτική συνοχή να είναι προσβάσιμη σε όλες τις περιοχές, ε, κυρίως αυτές που υστερούν περισσότερο, ε, για να έχουμε μια πιο ομαλή, μια πιο ισότιμη μετάβαση. Ποια, ποιοι είναι αυτοί οι τρεις βασικοί όροι που προανέφερα. Ε, είναι ε, που είναι απαραίτητη για να έχουμε μια αποτελεσματική μελλοντική πολιτική. Λοιπόν, η γεωγραφική κάλυψη της περιφερειακής πολιτικής, αυτό ε, εξαρτάται από την συνολική ικανότητα που έχουμε να πείσουμε τις εθνικές κυβερνήσεις και τους επικριτές ότι έχει αλλάξει η πολιτική για κάποια λίγα ε, κέρια σημασία ζητήματα που θα κρίνουν το μέλλον αυτής της πολιτικής. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον Φιλίπ Μάιστατ, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Επίσης θα ήθελα να πω ότι χωρίς τον Φιλίπ Μάιστατ τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής δεν θα κατάφερνε να περιλάβει καινοτόμες μεθόδους χρηματοδότησης. Σας ευχαριστώ θερμά, Φιλίπ, και εσάς και τους συνεργάτες σας. Πείτε, πείτε μας κάτι καλό για τα μελλοντικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ευχαριστώ, Ντανούτα. Κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, κυρία Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ της πατρίδας μου της Βαλονίας, της δικής μου περιφέρειας. Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά που με προσκαλέσατε και πάλι σε αυτή την έκδοση των ανοιχτών ημερών και χαίρομαι ιδιαίτερος γιατί η επιλογή του θέματος για τις φετινές ε, ανοιχτές μέρες είναι πολύ επίκαιρο γιατί η ανταγωνιστικότητα θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην επιτυχία της μελλοντική μας στρατηγικής της Ευρώπης του 2020. Η περιφερειακή ανάπτυξη ήταν μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων από την δημιουργία της το 1958 από τη Συνθήκη της Ρώμης. Και με βάση τη συνθήκη η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει ως αποστολή της την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Δηλαδή οφείλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία και προτεραιότητα σε προγράμματα και σχέδια που εκπορεύονται από τις ε, περιφέρειες της σύγκλησης, όπως λέμε. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στις δραστηριότητες των τελευταίων 50 χρόνων δεν ε, απομακρύθηκε ποτέ από αυτή την προτεραιότητα. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές εξακολουθούν να διαδραματίζουν και σήμερα το σημαντικότερο εταίρο μας ε, στις δραστηριότητες της ΕΤΕ και υποστηρίζουμε τις περιφερειακές και τοπικές αρχές είτε με άμεσο τρόπο, γιατί έχουμε άμεσες επαφές με τις περιφέρειες και τις πόλεις, αλλά και μέσω συγχρηματοδότησης των δραστηριοτήτων μας ε, και των δραστηριοτήτων τους, μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω παροχής τεχνικής αρρωγής και πρόσφατα με κάποιους τρόπους ε, δημοσιονομικών ε, διευκολύνσεων. Για παράδειγμα, την τελευταία τριετία, δηλαδή το 2007-2009, χρηματοδοτήσαμε δάνεια για κάποια σχέδια στις περιφέρειες ε, σύγκλησης για 66 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ε, ουσιαστικά το 40% του συνολικού όγκου ε, του δανεισμού. Και μάλιστα υπήρξε μια καλή ε, ισορροπία μεταξύ των 15 χωρών και των, των 12 χωρών πριν την πρώτη τελευταία διεύρυνση. Και μάλιστα μπορεί κατά κεφαλήν οι νέες χώρες να έχουν λάβει και περισσότερα κονδύλια και μεγαλύτερα δάνεια. Έχουμε πολλές κοινέ πρωτοβουλίες και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα όταν η κυρία Τανίτα Χιούμπνερ ήταν αρμόδια Επίτροπος Περιφερειακής ανάπτυξη. είχαμε αρκετέ τέτοιε κοινέ πρωτοβουλίε. Θα σα αναφέρω δύο το Jaspers, για παράδειγμα. Το Jaspers είναι ε, ένα μέσο τεχνικής ε, αρρωγής προκειμένου να βοηθήσουμε τα νέα κράτη-μέλη να προετοιμάσουν ε, μεγαλεπίβολα σχέδια υποδομής που θα χρηματοδοτούνται από τα Διευθυντικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Επίσης το Jessica που είναι μια κοινή πρωτοβουλία για την βοήθεια των ε, περιφερειακών αρχών προκειμένου να προβούν σε επενδύσεις ε, για την αηφόρο ανάπτυξη. Και η στρατηγική του 2020 δίνει κίνητρα και ενάυσματα καθώς και νέους προσανατολισμούς στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής και ταυτόχρονα αναγνωρίζει το νευραλγικό ρόλο που διαδραματίζουν οι περιφέρειες και οι πόλεις στην Ένωση. Δίνουμε έμφαση στην καινοτομία, την τεχνολογική ανάπτυξη, την φιλοπεριβαλλοντική ενέργεια. Υποστηρίζουμε την οικονομία της γνώσης και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με όλους αυτούς τους τρόπους προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών πόλων και περιφερειών. Έτσι προσπαθούμε να υλοποιήσουμε το στόχο για ε, ανάπτυξη που θα είναι έξυπνη, αηφόρο, αηφόρος και δεν θα αποκλεί κανέναν. Βέβαια η χρηματοδότηση καινοτόμων σχεδίων μπορεί να προσκρούσεις σε κολλήματα όπως η περιπλοκότητα των προϊόντων, τεχνολογικά προβλήματα, ε, δημοσιονομικές ή οικονομικές ε, δυσχέρειες που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια, κάποια προθυμία των τραπεζών, γιατί πολύ συχνά οι τράπεζες ε, δεν προσφέρονται να επενδύσουν σε άειλες, σε άειλες προτεραιότητες. Πάντως θεσμικά όργανα της Ένωσης όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αλλά και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να δημιουργήσουμε μια σειρά μηχανισμών που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Θα σας αναφέρω δύο από τα μέσα αυτά. Το Jeremy, για παράδειγμα. Το Jeremy είναι ένας μηχανισμός που δίνει την ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία και επιδοτήσεις Επίσης δημιουργούνται κάποια revolving funds για να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, σε δάνεια εγγύηση κτλ. Και υπάρχει και το RSFF, η χρηματοοικονομική διευκόλυνση για την επιμερισμό κινδύνου για την έρευνα. Είναι ένα κοινό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που επιτρέπει τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων και όπως σας είπα, αυτός ο μηχανισμός, αυτό το χρηματοοικονομικό μέσο είναι διαθέσιμο και στις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές. Ήδη μερικές περιφέρειες έχουν ε, αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα, γιατί το RSFF είναι προσιτό και σε τοπικές και περιφερειακές αρχές. Επίσης υπάρχουν και άλλα προϊόντα της ΕΤΕ που προβλέπονται στους τρεις πυλώνες του, της Ευρώπης το 2020, για παράδειγμα δάνεια για διαρθρωτικά προγράμματα που βοηθούν στην εφαρμογή των ε, προγραμμάτων διαρθρωτικών ταμείων και υποστηρίζει την ε, διαχείριση των επενδύσεων από τις περιφερειακές αρχές και μάλιστα συνεργαζόμαστε με τον Επίτροπο Χάν και το επιτελείο του προκειμένου να βελτιώσουμε την ε, αποτελεσματικότητα όλων αυτών των δημοσιονομικών και χρηματοοικονομικών εργαλείων. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ολοκληρώσω επιμένοντας σε ένα σημείο που κατά τη γνώμη μου είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Όπως ανέφεραν και οι προλαλήσαντες, η πολιτική συνοχής θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της νέας στρατηγικής Ευρώπη 2020. Και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η Στρατηγική Ευρώπη 2020 απαρτίζεται από τρεις πυλώνες. Σίγουρα χρειαζόμαστε την ευφυή ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε μια έξυπνη ανάπτυξη που θα επενδύει καλύτερα και περισσότερο σε έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και πληροφορία. Φυσικά χρειαζόμαστε και αηφόρο ανάπτυξη, μια βιώσιμη ανάπτυξη που θα σέβεται περισσότερο το περιβάλλον και που θα είναι πιο ε, λιτή στη χρήση των ε, φυσικών πόρων που θα πρέπει να αφήσουμε και τι επόμενε γενίε. Αλλά χρειαζόμαστε και μια ανάπτυξη που δεν θα περιθωριοποιεί κανέναν, δεν θα αφήνει κανέναν εκτό νυμφώνο και δεν θα αφήνει κανέναν πίσω στο δρόμο τη. Αν τα αποτελέσματα αυτή τη στρατηγική Ευρώπη 2020 ε, θα οδηγήσει στο να γίνουν πλουσιότεροι πλούσιοι και ισχυρότεροι ισχυροί, χωρίς ταυτόχρονα να βοηθήσει και τους φτωχούς να καρποθούν τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής, τότε μια τέτοια στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 θα είναι αποτυχημένη. Δεν θέλουμε καμία κοινωνική ομάδα και καμία περιφέρεια να μην μείνει στο περιθώριο και να μην ωφεληθεί από αυτή την ε, γενικότερη ανάπτυξη. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι αποφασισμένη να συμβάλλει με του μετόχου τη, τα κράτη-μέλη δηλαδή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε συνεργασία με τι τοπικέ και περιφερειακές αρχέ, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια πιο δυναμική ανάπτυξη αλλά και πιο ισορροπημένη ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωση. ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές μας και τώρα παραδίδω για την υπόλοιπη ε, συνεδρίαση το συντονισμό στο Μάρκ Ρότζερσον και ελπίζω να κάνει θαύματα και να σας ικανοποιήσει όλους το λίγο χρόνο που έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, όντως, κυρίες και κύριοι, τώρα έχει έρθει η ώρα της συζήτησης και των τοποθετήσεων. Ε, ε, ήδη έχουν ζητήσει το λόγο πολύ. Αν θέλετε να μιλήσετε, παρακαλείστε να ε, δώσετε το αντίστοιχο έντυπο στους κλητήρες. Δύο λεπτά έκαστος παρακαλώ ο μιλητής και να το σεβαστείτε. Τρεις προέδρους έχω, έναν αντιπρόεδρο, ένα επίτροπο ε, και ε, ένα πρόεδρο εδώ και όλοι θα σας παρακολουθούμε και θα φροντίζουμε να τηρείτε το δίλεπτό σας. Um, ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μίχαελ Σνάιντερ που εκπροσωπεί το Λαϊκό Κόμμα στην Επιτροπή Περιφερειών. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι πρόεδροι, κύριε επίτροπε, Αποτελεί χαρά για μένα να βρίσκομαι εδώ για 8 ε, φορά ε, στην εναρκτήρια συνεδρίαση των ανοιχτών ημερών με τις ε, πολλές διοργανώσεις, τα εργαστήρια, τα σεμινάρια. Φαίνεται πόσο μεγάλη και βαθιά είναι η προσήλωση των περιφερειών και των πόλεων της Ευρώπης για την Ευρώπη και πώς θέλουμε να συνεισφέρουμε για την Ευρώπη. Φέτος, το είπαν και οι προλαλήσαντες, το σύνθημα είναι η μελλοντική πολιτική συνοχή ε, ε, τη στρατηγική της Ευρώπης για το 2020. Στην Επιτροπή των Περιφερειών ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα εντατικά του περασμένου μήνε και καταλήξαμε όπως και πολλοί άλλοι ότι η στρατηγική της Λισαβόνας απέτυχε στους στόχου της ακριβώς γιατί δεν ε, συμπεριελάμβανε με τον τρόπο που του ήρμοζε και τι περιφέρειες και τι πόλει. Θα πρέπει λοιπόν να εξάγουμε τα διδάγματά μα. αλλά έχουμε αμφιβολίες αν κατά πόσο πραγματικά έχουμε βγάλει τα σωστά διδάγματα από την αποτυχία της Λισαβόνας. Η στρατηγική για το 2020 σε ό,τι αφορά το ρόλο των Δήμων και των Περιφερειών δεν αναφέρεται σχεδόν καθόλου σε αυτό. Στα κράτη-μέλη, στο βαθμό που μπορώ να το παρακολουθήσω, για την υλοποίηση της νέας στρατηγικής. Επίσης δεν έχει ξεκινήσει καν η συζήτηση για τη συμμετοχή των περιφερειών και των πόλεων και χάνουμε πολύτιμο χρόνο. Υπό την έννοια αυτή ε, είμαι πολύ ευγνώμων προς τη Βελγική Προεδρία που παρακάλεσε πριν από λίγους μήνες να κάνει έκθεση πρωτοβουλίας η Επιτροπή Περιφερειών για την Ευρώπη το 2020 και την πολιτική συνοχή. Αύριο θα συζητήσουμε την γνωμοδότηση αυτή και θα την εγκρίνουμε. Και για μας ε, είναι από τους σημαντικότερους ε, τομείς αυτούς και ε, ε, το θέμα των ε, εδαφικών συμφώνων. Δηλαδή, στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το κάθε επίπεδο. Τι ρόλος αναλογεί σε κάθε επίπεδο πολιτικής. Δεν θα πρέπει αυτά να τα αφήνουμε στην τύχη, αλλά να τα ορίζουμε και να τα καθορίζουμε. Από την άλλη, Έχουμε και τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα που είναι επίσης το σωστό πλαίσιο. Και ένα τρίτο, ε, η Επιτροπή Περιφερειών θα κάνει μια πλατφόρμα παρακολούθησης της στρατηγικής 2020 για να συνοδεύει σε επίπεδο θεσμικών οργάνων και στη συζήτηση της Βρυξέλλες και να μπορεί ε, να ε, κάνει τις προτάσεις της και να λέει πώς εφαρμόζεται αυτή η στρατηγική, πώς μπορεί να βελτιωθεί. Δύο λεπτά ακριβώς παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Σνάιντερ, όντως. Ισχυρή έκκληση για περιφερειακά σύμφωνα. Ακούσα ο κύριος Λάμπερντ Βανίστεροι, ε, συντονιστή ε, του ΕΛΚ της ε, Επιτροπής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Και από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σας καλωσορίζουμε θερμά στον οίκο της Δημοκρατίας, στο ημικύκλιο εδώ της Ολομέλειας. Έχω την εντύπωση ότι Καλά κάνουμε εδώ τη συζήτηση για τη συνοχή. Πριν από δύο χρόνια δεν ξέραμε τι ήταν η συνοχή. Ένα non-paper το είχαν παραγωνίσει κάπως και τώρα ίσως και χάρη στην κρίση ερχόμαστε στα θεμελιώδη. Τέσσερις παρατηρήσεις έχω ε, σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Σνάιντερ. Συμμετοχή των περιφερειών και των πόλεων στην Ευρώπη του 2020, στη στρατηγική αν διαβάσετε τα κείμενα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που συνεργάζονται, αλλά δεν εφαρμόζουν την επικουρικότητα. Και το Περιφερειακό Σύμφωνο ή το Σύμφωνο της Εδαφικής Συνεργασίας είναι πραγματικά κάτι που πρέπει να οριστεί και το συζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεύτερον, σε όλη την επικράτεια δεν ισχύει αυτό. Υπάρχουν ακόμα περιφέρειες και πόλεις που νομίζουν ότι μπορούν να είναι κάποιες λευκές ε, περιφέρειες από πλευράς ανταγωνιστικότητας, απασχόλησης. Όχι, η συνοχή καλύπτει το σύνολο της επικράτειας, αλλιώς είναι λάθος. Και ε, ακούστηκε και ε, η εδαφική συνοχή, όχι οι πλούσιοι να γίνουν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι και να μένουν πίσω. Τρίτον, τα λεφτά. εδώ είναι το θέμα, το οικονομικό χρηματοδότηση. Ε, είτε είναι ενεργειακό ταμείο, κλιματικό ταμείο, ε, ε, ταμείο υδάτων, ξέρω εγώ, είπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι. Θα πρέπει να είναι οριζόντια η ενίσχυση των περιφέρειων. Και τέταρτον, δεν είστε μόνο εδώ αυτή τη στιγμή δική μας προσκεκλημένοι. Ε, υπάρχει Επιτροπή Περιφερειών με την Επιτροπή της που ονομάζεται ΚΟΤΕΡ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση και αυτό είναι στο ίδιο επίπεδο τώρα το Κοινοβούλιο, 100% συναπόφαση και να απευθύνεστε σε εμά πάντοτε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε πίσω στην Επιτροπή των Περιφερειών τώρα. Καρλ Χάιντς Κλέρ, πρόεδρος των Σοσιαλιστών στην Επιτροπή των Περιφερειών. Παρακαλώ. Thank you. Acting chair. Ευχαριστώ. Όταν ήρθα στην Επιτροπή Περιφερειών πριν από 15 χρόνια, με ρώτησε ο καλύτερος μου φίλο, μα γιατί το κάνεις αυτό, γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου, Βρυξέλλες, τώρα Ευρωπαϊκή Ένωση, πού πας εκεί. Και το απάντησα διότι την Ευρωπαϊκή Ένωση το θεωρώ το μεγαλύτερο πολιτικό επίτευγμα του 20ου αιώνα. Μετά από δύο πολέμους, παγκοσμίους παρακαλώ, με τρομακτικά δεινά, ατελείωτα, οι ιδρυτές, οι πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να συνεργαστούν. Όχι πια ε, πολεμικές ε, σειράξεις, αλλά συνεργασία. Με στόχο μια πιο στενή ένωση των λαών. Λοιπόν, συνοχή στην Ευρώπη. Και Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία πολιτική που να είναι πιο σημαντική για αυτό το στόχο. Είναι η πολιτική συνοχή και η περιφερειακή πολιτική, την οποία εκπροσωπεί ο Επίτροπο κ. Χάν. Είναι η σημαντικότερη πολιτική για τη συνοχή τη Ευρώπη. Και ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική όσο του σημερινού καιρού τη κρίση που ζούμε. Διότι είναι αλήθεια αυτό. Είμαστε στην πιο σκληρή και οξία κρίση που έχουμε ζήσει ποτέ. Η πόλη αυτή των Βρυξελών θα πρέπει να προσέξει να μην γίνει Washington DC χωρίς το Tea Party γύρω γύρω. Εκεί όμως το πάμε, προς τα εκεί οδεύουμε. Κοιτάξτε πώς συμπεριφέρονται οι λαοί της Ευρώπης. Τι πιστεύει ο κόσμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Πάρα πολύ επικριτικά και κρίσιμο αυτό. Το ίδιο συμβαίνει στις ΗΠΑ με τη Washington. Αν θέλουμε να τα αλλάξουμε αυτό ξανά, τότε θα πρέπει να έχουμε μια πολιτική που να ενισχύει πραγματικά και να προωθεί τη συνοχή και να είναι μια πολιτική κατά της χρηματοπιστωτικής κρίσης και κατά της οικονομικής κρίσης που παραμένει έχουμε τη μεγαλύτερη ανεργία από το 1999 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να είναι λέω μια πολιτική η οποία να μην υπηρετεί μόνο τους έχοντες και κατέχοντες, αλλά και τους φτωχούς και τα μεσαία στρώματα και τους απασχολούμενους. Αυτό χρειάζεται. Και ε, απαιτείται ε, άμεσα να γίνει αυτό. Και αν το καταφέρουμε αυτό, ο πρόεδρος... Ε, τελειώνω. Ε, για να ανέβει και το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μάτια του πληθυσμού. Είναι καλή ευκαιρία λοιπόν οι νυχτέ ημέρε να ε, προχωρήσουμε σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Um, uh, ευχαριστώ. Επιστρέφουμε τώρα και πάλι στην ε, Επιτροπή Περιφερειακής Αναπτύξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, Ρικάρντο Κόντες Λάστρα. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητήσουμε εδώ όλοι μαζί στο πιο σημαντικό φόρουμ της Ευρώπης. Γιατί στο φόρουμ αυτό όλες οι περιφέρειες ανταλλάσσουμε τις ιδέες μας και συμμεριζόμαστε το κοινό αυτό όραμα. Γι' αυτό θα ήθελα να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να διατρανώσω τη σημασία της πολιτικής συνοχής για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Ο μελλοντικός λοιπόν προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να θεωρεί την πολιτική συνοχή ως πολιτική ανάπτυξης και όχι πολιτική δαπανών και εξόδων. Όλοι πιστεύουμε ότι η πολιτική συνοχή διευκολύνει τον εξυγχρονισμό και την βιώσιμη ανάπτυξη και δείχνει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη γιατί έχει επιρροή στην απασχόληση, την έρευνα, την καινοτομία, τις μεταφορές, τις κλιματικές αλλαγές, τις υποδομές, την ενέργεια, την καταπολέμηση της ένδυας. Όλα αυτά τα θέματα είναι κεφαλαιόδου σημασία για την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρί την ανάμειξη των ευρωπαϊκών περιφερειών. Γιατί οι περιφέρειε βρίσκονται κοντά στον πολίτη. Αυτέ βρίσκονται στο πλευρό του. Και οι ευρωπαϊκέ περιφέρειε είναι αυτέ που μπορούν να κάνουν το μέσο στην ε, κοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε προασπίσουμε την πολιτική συνοχή ω σημαντική ευρωπαϊκή πολιτική και να μην ενδώσουμε στον πειρασμό τη επανεθνικοποίησής τη, Όχι μόνο για την απήχηση που θα έχει στην ανάπτυξη των περιφερειών και των κρατών μα, γιατί η πολιτική συνοχή έχει προστιθέμενη αξία σε αυτή την δύσκολη οικονομική εποχή που διανύουμε. Γιατί η πολιτική συνοχή δίνει ορατότητα και προβολή στην ευρωπαϊκή πολιτική και είναι ε, από του ακρογωνιού λίθους τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Επίσης θα πρέπει να μην ξεχνούμε τον κεφαλαιόδη ρόλο που παίζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες, αλλά ταυτόχρονα να μην ξεχνούμε και το σημαντικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Μία αποκεντρωμένη διαχείριση και μία πολυεπίπεδη διακυβέρνηση είναι κλειδιά για να εξασφαλίσουν την επιτυχία της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Thank you Um, σας ευχαριστώ. Τώρα θα ακούσουμε τον Πρόεδρο των Φιλελευθένων της Επιτροπής των Περιφερειών, Φλό Κλούκλας, που ανήκει και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Λίβερπουλ. Um, ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να σας ε, χαιρετήσω εξ ονόματος της Ομάδας των Φιλελευθένων της Επιτροπής των Περιφερειών. Η πέμπτη έκθεση συνοχής ακόμη δεν έχει δημοσιευθεί αλλά ε, έχουν, ε, υπάρχουν εικασίε πολλέ για το περιεχόμενο. Κάποιοι ξέρουν τι λένε, κάποιοι ίσως λιγότερο. Ε, τώρα, αυτοί που ξέρουν, γνωρίζουν τα πράγματα και έχουν κάνει τις παρατηρήσεις τους για την επικείμενη έκθεση συνοχής, αν έχουν δίκιο, τότε θα συμφωνήσει η Επιτροπή των Περιφερειών και θα συμφωνήσουν και πολλές πόλεις και πολλές περιφέρειες στα κράτη-μέλη. Χάρηκα ιδιαίτερα στον άκουσα το μήνυμα του Πρόεδρου Μπαρόσο. Είπε ότι οι βασικέ αρχέ ε, τη πολιτική συνοχή ε, που θα σκιαγραφούνται σε αυτή την πέμπτη έκθεση ε, θα παραμείνουν αναλύωτε. Όλοι γνωρίζουμε, Φερρυπίν, ότι οι μεταβατικές περιοχές θα συμπεριληφθούν σε οποιασδήποτε συζητήσεις γίνουν και πολλές από αυτές τις περιοχές που ανήκουν στο λεγόμενο phasing in, που εισέρχονται τώρα δηλαδή στη μεταβατική φάση, θα καλυφθούν επίσης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Κάποιες από αυτές τις περιοχές ε, πρέπει να τις χειριστούμε τώρα γιατί έχουν δυσκολίες ε, διότι ε, δεν μπόρεσαν να τραβήξουν άλλο δαπές επενδύσεις από τον περασμένο Ιανουάριο και άρα θα, αυτό θα πλήξει τις επιχειρήσεις. Ελπίζω λοιπόν να ρυθμιστεί αυτό το ζήτημα με την πέμπτη έκθεση. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Εάν θέλουμε μια πολιτική συνοχή που όπως είπατε και εσείς δεν μοιράζει απλώς κονδύλια αλλά βοηθάει, τονώνει την ανάπτυξη πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, διαλλακτικοί και να επικουρούμε τις περιοχές όταν και όπου το χρειάζονται. Και για ποιο λόγο είναι πάρα πολύ απλό. Χρειαζόμαστε θέσεις εργασίας για τους πολίτες, χρειαζόμαστε ανάπτυξη για την οικονομία μα οι θέσει απασχόλησης και η οικονομία. Ή πρέπει αυτή να είναι ε, η δίδυμη στόχη της πολιτικής. Για να τελεσφορήσει η πολιτική, τι θα κάνουμε όμως. Ε? Ε, η συνθήκη, η στρατηγική της Λισαβόνας δεν τελεσφόρησε γιατί δεν είχε ιδιοκτήτη. Και τώρα ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες όλοι, οι πόλεις, τα χωριά, τα κράτη-μέλη. Αν θέλετε να επιτύχει η Ευρώπη 2020 την ιδιοκτησία, την νομή θα πρέπει να την έχουν όσοι ζουν εκεί, όσοι κυβερνούν εκεί, όσοι εργάζονται εκεί και όχι απομονωμένοι γιατί και οι πολίτες ε, πρέπει να εμπλακούν στη διαδικασία και είχαμε και νωρίτερα φέτος ε, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Συμμετοχή των Πολίων και τονίστηκε αυτό γιατί, διότι Επίτροπε, κύριε, ε, σας παρακαλώ να είστε σύντομοι διακόπτεται η ομιλήτρια, διότι η πολιτική συνοχή είναι το πρόσωπο της Ευρώπης στις περιφέρειές μας, στις πόλεις μας. Ε, χωρίς αυτό θα ε, εκλείψει η Ευρώπη. Οι πολίτες πια δεν θα ξέρουν τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για αυτούς τους ίδιους, γι' αυτό και σας ζητώ ε, να σκεφτείτε πώς ακριβώς, ε, με ποιο τρόπο οι χώρες μας, οι πόλεις, οι υπεθρός μας, όλοι πώς θα συμμετάσχουν σε αυτή την πολιτική έχοντας κατά νου αυτό που λέμε στη δικιά μου την περιοχή και ελπίζω να το δεχτείτε, ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Ε, αυτά θα βοηθήσουν και θα βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο λόγια, αν και ήταν πάνω από δύο λεπτά, εν πάση περιπτώσει. Και τώρα... Ο κύριος Γέρση Ζακά, πρόεδρος της ομάδας του στην Επιτροπή Περιφερειών. Ευχαριστώ. Αξιότιμα μέλη του Προεδρείου, η σημερινή σύνοδος είναι πολύ σημαντική και θα ήθελα να σε απευθύνω το χαιρετισμό τη ε, ομάδα του συνασπισμού. Η στρατηγική τη Ευρώπη του 2020 θα επηρεάσει και την οικονομική και την κοινωνική κατάσταση ολόκληρη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά, η αποτελεσματικότητά τη θα εξαρτηθεί από την ενεργό ανάμειξη όλων των σημαντικών ενδιαφερομένων στην υλοποίηση των στόχων τη Στρατηγική του 2020. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμμεριστούν τους στόχους και να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην υλοποίησή τους. Το βασικό στοιχείο της στρατηγικής του 2020 θα πρέπει να εξακολουθήσει να παραμείνει η εδαφική συνοχής που έχει κατοχυρωθεί πλέον και στη συνθήκη της Λισαβόνας και στη στρατηγική της Λισαβόνας. Κάτι τέτοιο προποθέτει φυσικά ανάμειξη σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνηση κάθε ευρωπαϊκή πολιτική σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό είναι και τοπική πολιτική και περιφερειακή πολιτική. Γι' αυτό και η συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην ανάπτυξη, στη χάραξη και την εφαρμογή μια τέτοια στρατηγική είναι απαραίτητη και θα έλεγα κεφαλαιότου σημασία. Επίση, ε, σημαντική είναι και η οικονομική συνοχή. Γιατί με την οικονομική ανάπτυξη θα καταφέρουν όλε οι περιφέρειέ μα, οι δήμοι, οι κοινότητε και όχι μόνο οι πόλει χάρη στην αξιοποίηση των πόρων και της τεχνογνωσίας μπορούμε να φτάσουμε στο, στην πλήρη αξιοποίηση του οικονομικού δυναμικού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτύχει και οι στόχοι της θα υλοποιηθούν μόνο αν τους καρπούς της τους απολαύσουν όλες οι, όλες οι περιφέρειες και όλες οι δήμοι και όλοι οι Δήμοι. Θα πρέπει να μην ε, συγκεντρώσουμε τους στόχους μόνο στις πόλεις και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Θα πρέπει τα κονδύλια να φτάσουν σε όλες τις περιφέρειες και περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και την γεωργία και την πολιτική των τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τη διαμόρφωση αυτών των πολιτικών. Και μας, ε, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα στις τοπικές και περιφερειακές αρχές το θέμα και της ανάπτυξη τη υπαίθρου Οπότε όλες οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα πρέπει να μελούν και την ανάγκη ανάπτυξης της υπαίθρου και την ανάπτυξη της γεωργίας. Γιατί περίπου 30 ε, εκατομμύρια άνθρωποι απασχολούνται στη γεωργία και 40 εκατομμύρια στην ε, βιομηχανία τροφίμων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το θέμα. Η πολιτική συνοχή λοιπόν θα πρέπει να λάβει υπόψη και την κατάσταση των κατοίκων της υπαίθρου. Ευχαριστώ. Uh, Σας ευχαριστώ. Επανερχόμεθα στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάριν Κάντεμπαχ ε, θα πάρει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και συγχαρητήρια για τη σημερινή διοργάνωση, ε, την 8η. Εγώ είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μόλις εδώ και ένα χρόνο αλλά γνωρίζω τις Open Days από χρόνια γιατί ήμουνα 16 χρόνια στην περιφερειακή ε, αυτοδιοίκηση, στην τοπική, 7 χρόνια στην περιφερειακή, ε, σε τοπικά κοινοβούλια και είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργάζονται αυτά τα επίπεδα. Σε όλα τα πολιτικά επίπεδα θα πρέπει να φροντίζουμε για ποιότητα ζωής και ε, το άμεσο περιβάλλον των ανθρώπων είναι οι δήμοι και οι κοινότητες και μετά οι περιφέρειες αν δεν είναι ε, καλή η ποιότητα ζωής τόπου, όσο καλά και να τα λένε οι ευρωπαϊκές στατιστικές, ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος. Χρειάζεται λοιπόν μια πολιτική συνοχής και είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί έχει τρεις σημαντικές αποστολές. Πρώτον, ποιότητα ζωής και ανταγωνιστικότητα όμως στην Ευρώπη και στην επικοινωνία θα πρέπει να το τονίζουμε πολύ περισσότερο ότι τα χρήματα εκείνα που πηγαίνουν στην πολιτική συνοχής δεν είναι δωρεές σε οτιδήποτε περιφέρειες, έτσι γενικά το είπε και στην ακρόαση του Επίτροπος κύριος ε, Χάνα, μας είπε ότι είναι ο πατέρας των περιφερειών, ας είναι, αλλά θα πρέπει να πηγαίνουν τα χρήματα εκεί που πιάνουν τόπο, εκεί που ενισχύονται τα ταλέντα και η δημιουργικότητα. Χρειάζονται ένα έναυσμα και οικονομικό για να αναπτυχθούν οι περιφέρειες. Θα πρέπει να προσέχουμε ε, ε, όμως και οι ε, ανεπτυγμένες περιφέρειες να μην υποβαθμιστούν. Και το τρίτο είναι η Ευρώπη θα πρέπει να γίνει χειροπιαστή πραγματικότητα, κυρίως στις περιφέρειες, για να δείχνουμε στον ε, κόσμο επιτόπου πού πηγαίνουν τα κονδύλια για την εκπαίδευση, για την απασχόληση. Τότε θα είναι και πρόθυμοι να χρηματοδοτούν από κοινού την Ευρώπη. Γιατί χρειαζόμαστε και ε, πόρους και τα κράτη-μέλη στο Διενικές για να δίνουν αυτά τα χρήματα ε, θα ε, πρέπει να μπορούν να εξηγούν στους πολίτες πού είναι η προστιθέμενη αξία. Κάθε επιτυχία λοιπόν για τα 130 εργαστήρια και πιστεύω ότι θα είναι θαυμάσια η εβδομάδα που διανύουμε. Thank you very much indeed. Σας ευχαριστούμε. Δεν χρειάστηκε καν να πιάσω το σφυράκι μου. Ένα μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου της περιοχής Ουσίμα στο Ελσίνκι, Μάρκο Μακούλα, θα πάρει το λόγο. Arvoisa ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η πολιτική συνοχής ε, βασίζεται στην ε, συνεργασία ανάμεσα στις περιοχές αλλά και στο θάρρος, το κουράγιο των περιοχών να στραφούν στην καινοτομία. Βέβαια, υπάρχει το γνωστό χάσμα, μεγάλο χάσμα ανάμεσα στη θεωρία και στην πραγματικότητα. Ε, ακούσαμε διάφορες απόψεις, ε, πολιτικές ε, τοποθετήσεις, αλλά καλό θα ήταν να περάσουμε και σε κάποια πρακτικά στοιχεία, ε, μεριμνώντας ώστε να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο η, στρατηγική Ευρώπη 2020 για να έχουμε ένα νέο όπλο στα χέρια μας. Ε, έχουμε ήδη πολυάριθμες ε, ε, καλές πρακτικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από διάφορες γωνιές της Ευρώπης. Ο Επίτροπος Χάν μας κοινοποίησε το όραμα του για την πολιτική συνοχή και την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. Δεν χρειάζεται να είναι όλοι καινοτόμοι, δεν χρειάζεται όλοι να εμπλέκονται σε ερευνητικά προγράμματα. Το σημαντικό είναι τα αποτελέσματα της έρευνας να έχουν μια πρακτική έκφανση κάποια στιγμή. Χρειάζεται βέβαια συνεργασία ανάμεσα στις πόλεις για να έχουμε την κρίσιμη μάζα η οποία θα μας επιτρέψει στην Ευρώπη να ε, είμαστε πόλος έλξης ε, για τις επενδύσεις, ε, κυρίως για τις καινοτομίες και δει τις πλέον ριζοσπαστικές καινοτομίες. Έχουμε ήδη παραδείγματα ευφυής, μεταφορές, εφαρμοσμένη έρευνα, ε, αλλά δεν χρειάζεται κάτι ριζοσπαστικό, θέλω να πω. Έχουμε ήδη μέσα στη διάθεσή μας. Thank you very much indeed. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ακούσαμε τον Νότο. Όχι, πάμε στο... Πήγαμε από το... Πάμε, από, α, πάμε προς τον Νότο, πάμε από το Ελσίνκι στη Δουλκέρκη, ο κύριος ε, Μισελ Τελπά. Κυρίες και κύριοι, ε, αν ξαναρχίσω θα, ε, θα απευθυνθώ πάλι στις πρόεδρες. Συμφωνούν οι πάντες, οι πάντες. Εδώ στο παρόνιμη κύκλο οι πάντες συμφωνούν για την πολιτική συνοχή, για την ε, διακυβέρνηση σε πολλά επίπεδα, για το ρόλο των ΟΤΑ. Ήμουν κύριε Ντεμότ προχθές στο τουρνέ για να γιορτάσουμε ε, την 20η επέτειο του Ιντερεκ και όλοι ομόφωνοι για το ρόλο ε, των ε, περιφερειών και των τοπικών αυτοδιοικήσεων και τα 20 τελευταία χρόνια και εγώ είμαι ικανοποιημένο. Ευχαριστημένοι όλοι στη γυάλα μα. Απ' έξω τι γίνεται όμω. Εγώ γνωρίζω επιτρόπους που έχουν μία ιδέα. Να, να πάρουν τα λεφτά του Επιτρόπου Χάν. Και ξέρω και κυβερνήσεις που έχουν μία έμονη ιδέα να επανεθνικοποιήσουν τις πολιτικές. Ε, λοιπόν, αυτό που κάνουμε εμείς εδώ θα πρέπει να βγει και έξω από τη γυάλα και έξω από το ημικύκλιο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλη την Ένωση πρέπει να πείσουμε, όχι τους εαυτούς μας. Από την αρχή της συζήτησης συμφωνούσα με τα όσα έλεγαν οι συνάδελφοι του ΕΛΚ. Καταλαβαίνετε, άκουσον άκουσον πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Γιατί ζούμε την πραγματικότητα. Η αυριανή Ευρώπη ε, στις δικές μας επικράτησεις και στα εδάφη μας χτίζεται. Ε, εάν είναι αύριο η Ευρώπη δημοκρατική, αυτό θα γίνει γιατί θα έχουν δει επιτόπου τα αποτελέσματα οι δικοί μας πολίτες. Μια απλή παρατήρηση. Ας αξιοποιήσουμε τις ανοιχτές μέρες για να απευθυνθούμε προς τα έξω, γιατί είναι πάρα πολύ εκείνοι που θα πρέπει να πείσουμε έξω πολύ περισσότερο από τους εδώ παρόντες. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και καλό μας κουράγιο σε όλους μας. Thank you very much indeed. Σας ευχαριστώ. Σας διαβεβαίω πάντως ότι οι τρεις επόμενοι ομιλητές μας βρίσκονται εκτός ε, των της Πομφόλιγας των Βρυξελών. Από την Ιταλία, ο κύριος Μάσιμο Μπέλο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι ανοιχτέ αυτές οι μέρες είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία για τις ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες της Ευρώπης. Και από αυτή την άποψη θεωρώ ότι οι ευρωπαϊκές πόλεις αποτελούν το βασικό σημείο αναφοράς για τι συμβάλλουν και εδραιώνουν την ευρωπαϊκή πολιτική και στις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Και μάλιστα ήταν πολύ αξιόλογες ε, πολλές πρωτοβουλίες που αναλύθηκαν και τις αξιολογώ και τις, και ε, εκτίμησα ιδιαίτερα ως δήμαρχος, γιατί είχαμε μια πρωτοβουλία για την αηφόρο, ανα, αηφόρο ενέργεια και μάλιστα θυμάμαι ότι στις 4 Μαΐου υπογράψαμε εδώ στο ημικύκλιο επίσημα αυτή την πρωτοβουλία για την αηφόρο ενέργεια. Και θα ήθελα να απευθύνω μια πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν μπορούμε να διανοηθούμε ένα σύμφωνο, το, δεν μπορούμε να σκεφτούμε ένα σύμφωνο των δημάρχων για την πολιτική συνοχής, που θα είναι ένα σύμφωνο ευθύνη και ενεργού συμμετοχής όλων των πόλεων που θα εκπροσωπούνται από του Δημάρχου του, Γιατί μιλούσα, μιλήσαμε για τις περιφέρειες, αλλά και οι κοινότητε, και οι δήμοι είναι σημαντικό στοιχείο και απαραίτητο σημείο αναφορά τη Ευρώπη. Ο ευρωπαϊκό προπολογισμό θα πρέπει να είναι εργαλείο όχι μόνο κοινωνική αλληλεγγύη, αλλά ένα πολύ σημαντικό οικονομικό μέσο. Και μάλιστα η πολιτική μετά το 2013 ε, θα, θα πρέπει να υποτιμηθεί. Και οι δήμικοι κοινότητε λοιπόν θα μπορέσουν να πρωταγωνιστήσουν και στην περίοδο μετά το 2013. Και αν υπάρχουν κάποια προβλήματα, και θα ήθελα εδώ να ολοκληρώσω, γιατί θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες, πιστεύω ότι μπορούμε να μετατρέψουμε τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουμε σε ευκαιρίε. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο σε έναν καλεσμένο μας από τις Ηνωμένε Πολιτείε, τον καθηγητή Άντριαν Πατρέσκου, που είναι καθηγητής ε, στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ στις Ηνωμένε Πολιτείε. Έχετε το λόγο κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ. Πολύ ευγενικό εκ μέρου σα. Ευχαριστώ όλου του προέδρου, αντιπροέδρου και όλου του υπόλοιπου. Εγώ είμαι από το Πανεπιστήμιο τη Μέριλαντ. Διδάσκω και στη Γερμανία και στη Ρουμανία. Ε, ξέρετε ότι το όνομά μου έρχεται από την Κούνζοβα στα νότια του Δουνάβεως, ε, από τη, στη Βουλγαρία. Ε, και μου είπε η κόρη μου κάποια στιγμή, εγώ είμαι από παντού, από ολόκληρο τον κόσμο. Έξι ήταν τότε και μετά ακολούθησε ένας κατάλογος χωρών και πόλων με τις οποίες είχε κάποια σχέση. Η θρησκεία μου πια είναι, να κάνω το καλό. Το, ο Τόμας Πέιν το είπε αυτό ε, το, στο 1776, πριν την Τετάρτη Ιουλίου για την Ανεξαρτησία. Καταπληκτική, δεν καταπληκτική πρωτοβουλία, αλλά ε, θυμίζω ότι οι περιφέρειες είναι περίπλοκα συστήματα, άρα οι πρωτοβουλίες ε, που εκπορεύονται από αυτές ε, θα καταφέρουν να περάσουν ε, σίγουρα παρά τους φραγμούς που εμείς ορθώνουμε μπροστά τους. Πρέπει να άρουμε αυτούς τους φραγμούς, αυτά τα εμπόδια. Πολύ χαίρομαι, πολύ μιλάνε για πρωτοβουλίες από τη ρίζα προς τα πάνω. Άλλοι λένε να βγούμε από τη φυσαλίδα των Βρυξελών. Εγώ τα επικροτώ αυτά, χαίρομαι, αλλά ε, σας προτείνω ένα πολύ απλό πείραμα. Πριν από 30 χρόνια ήμουν 15 χρονών και πρότεινα στο διευθυντή του σχολείου μου το εξής να γίνονται εμπειρίες με την πράσινη τεχνολογία στο μάθημα της φυσικής. Είπε ο διευθυντής, ε, δεν μπορούμε, δεν είναι στη διδακτική ύλη σήμερα. Ζω στην Αμύρ κοντά στις Βρυξέλλες και ξέρω ότι πολλά παιδιά στο γυμνάσιο τους ρωτάω Ξέρετε τίποτα για πράσινες τεχνολογίες, σας μαθαίνουν τίποτα στο γυμνάσιο. Όχι μου απαντάνε τίποτα, μηδέν. Στο σχολείο κανείς δεν έχει μάθει ότι μπορεί να προκύψει ενέργεια από τον ήλιο. Ε, στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, έτσι, στο γυμνάσιο. Αυτά γίνονται στο πραγματικό κόσμο και ε, μπορεί... Θέλω να προτείνω τρία πράγματα. Γρήγορα να τα προτείνετε όμως, λέει ο συντονιστή. Ε, ε, θέλουμε... Ε, Ε, θέλουμε ένα σύστημα εθνικών πάρκων ε, για που θα συντονίζει όλα τα εθνικά πάρκα σε όλες τις χώρες. Επίσης, σε παιδικά μουσεία ε, για αυτούς που θα έχουν τις δουλειές, τις καινούργιες το 2020 για να είναι δημιουργικοί. Και τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό να γίνεται, γίνονται εκ περιτροπής οι συναντήσεις, δηλαδή να πάμε στην Κένζοβα, στη Βουλγαρία, την ε, όλοι μαζί την επόμενη φορά για να καταλάβουν και οι άνθρωποι εκεί ότι για αυτούς μιλάμε και για αυτούς αγωνιζόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much. Um, Σας ευχαριστούμε. Ε, θα είμαι ακριβοδίκαιος ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Περνάω τώρα στην ε, Ακαδημία Επιστημών της Μόσχας μετά τη Μέρλεντ. Ο, ο καθηγητής Σεργέη ο Ελπίζω να παραφθείρω το όνομά σα. Πάρα πολύ ωραία το προφέρετε. Ωραία. Στην ε, Ρωσία συζητούμε επιμακρών το κατά πόσο εμεί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική ή όχι. Βέβαια οι απαντήσεις ε, ε, ποικίλουν. Αλλά θα πρέπει να διδαχθούμε από τι εμπειρίε, όχι μόνο τι θετικέ, αλλά και τι αρνητικέ. γιατί οποιαδήποτε εμπειρία έχει κάποια ωφέλη γιατί η περιφερειακή πολιτική είναι μακροχρόνια πολιτική. Και τελικά η περιφερειακή πολιτική είναι μια ανεξάρτητη πολιτική από την εξωτερική πολιτική, την οικονομική πολιτική κτλ. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και το επιστημονικό έργο. Και θα πρέπει να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας. Έχουμε καλούς εμπειρογνώμονες. Θα πρέπει καταρχήν να ξεκινήσουμε από περιφερειακό, τοπικό, εθνικό επίπεδο και μετά να ανέλθουμε σε κεντρικό επίπεδο. Νομίζω ότι η εμπειρία των Δήμων είναι πολύτιμη και θα πρέπει να την ακούσουμε. Επίσης, θα πρέπει να αλλάξουμε και την ονομασία ανοιχτέ μέρε. Τι σημαίνει ότι οι ανοιχτέ μέρε είναι μόνο αυτέ οι πέντε μέρε και όλε οι υπόλοιπε μέρε είναι κλειστέ μέρε. Να μιλάμε για ανοιχτά χρόνια. Να μην μιλάμε για ανοιχτέ μέρε μόνο. Ευχαριστώ. Ναι, καλό είναι να βγούμε από τη φυσαλίδα ή τη γέρα των Βρυξελών. Στο κάτω-κάτω είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσκεκτημένοι του Κοινοβουλίου. Οπότε ζώσουμε δώσουμε το λόγο τώρα σε ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την ομάδα των φιλελευθέρων, ο Μάικλ Τιούρερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Πολλά υπόθηκαν ήδη για τη διαρθρωτική πολιτική και την πολιτική συνοχή. Νομίζω ότι μα περιμένουν μεγάλε αποστολέ. Η κρίση του ευρώ, η κρίση των κρατικών χρεών φτάνει ε, στους πολίτες μας. Και ποιον αντιμετωπίζουν οι πολίτες, τα ξέρω εγώ ως δήμαρχος και ως μέλος Περιφερειακού Κοινοβουλίου, στις περιφέρειες και περισσότερο από ποτέ θα πρέπει να ενισχύσουμε την πολιτική συνοχή και τη διαρθρωτική πολιτική και να συζητήσουμε ακριβώς τι προσφέρει η πολιτική αυτή για την υπέρβαση της κρίσης αυτής. Τι προσφέρει και πώς συνεισφέρει στη μακροοικονομική σταθεροποίηση και εδώ έρχεται το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας στο επίκεντρο. Θα πρέπει ακριβώς αυτό να εστιάσουμε γιατί το ταμείο είναι μείον. Γιατί θα πρέπει η διαρθρωτική πολιτική και η συνοχή να αρχίζει στη ρίζα του κακού, στη δημιουργία του θέσεων απασχόλησης, στο να λειτουργούν οι υποδομές. Και εκεί έρχονται ε, στο επίκεντρο μικρομεσα... οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το 99% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη είναι μικρομεσαίες. Αλλά μόλις το 8% συμμετέχει στην εσωτερική αγορά. Γι' αυτό εμείς ως φιλελεύθεροι ζητούμε ένα νέο προσανατολισμό της πολιτικής αυτής που να λαμβάνει σοβαρά υπόψη ε, τις περιφέρειες που κάνουν προσπάθειες να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα, μεταφορά τεχνογνωσίας, εφαρμοσμένη έρευνα ε, στην πραγματικότητα, βεβαίως και γέφυρες με τα πανεπιστήμια αριστείας και ικανότητας για να αναπτυχθούν οι περιφέρειες μας και να βοηθήσουμε ακριβώς εκείνες τις περιφέρειες που χρειάζονται περισσότερη βοήθεια. Και υπάρχουν στρατηγικές μακροπεριφερειών της Βαλτικής ή του Δουνάβεως ή ε, του Ευξήνου Πόντου. Ευχαριστώ. Thank you very much Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο για να μιλήσει μάλιστα η κυρία εκεί πίσω με το Τυρκουάζ. Μπορείτε να συστηθείτε. Μαρτίν Τεβενιό από τη Γαλλία και εκπροσωπώ ένα δίκτυο που ονομάζεται Δίκτυο Περιφερειακών Τοπικών Συμφώνων. Είμαστε πεπισμένοι ότι χρειάζεται να ξεκινήσουμε και πάλι από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή, ε, επί τόπου ε, λύνονται τα προβλήματα, δίνονται ε, οι λύσει σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Έτσι οργανώνεται η λύση. Έχω την αίσθηση ότι εδώ εκπροσωπώ την κοινωνία των πολιτών και θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, μάθουμε να συνεργαζόμαστε με την κοινωνία των πολιτών αντί να μιλάμε για την κοινωνία των πολιτών. Και χαίρομαι που ε, έχει με μέρημνα για το θέμα αυτό και θα συζητήσουμε και την κοινή δράση και την κοινή ευθύνη μας και πώς από κοινού θα βρούμε κάποια στοιχεία ή κάποιες απαντήσεις για να τα εντάξουμε σε λύσεις απτές, χειροπιαστές. Οι πολίτες θα μπορούν να επαληθεύουν εάν τα όσα πρότεινα, τα όσα είπαν, ελήφθησαν υπόψη σε κάποιες λύσεις που ορισμένοι τους προσφέρουν έξωθεν. Αυτή λοιπόν είναι μια διαδικασία εκμάθησης της κοινή ευθύνη, της κοινή μοίρα μαζί με τους πολίτες γιατί τόπου βοηθούν πολύ οι πολίτες. Thank you very much. Any... Σας ευχαριστώ. Έχει περισσέψει λίγος χρόνος. Αν θέλει κανείς το λόγο μπορεί σύντομα να τον λάβει. Επαναλαμβάνω, θέλει κανείς το λόγο, το κρατήριο. Χέρι είναι αυτό που βλέπω. Μάλιστα. Η κυρία με τα μαύρα στο έδρανο 484. Ευχαριστώ. Ονομάζομαι ε, Τζόζεφι Ραμπόλα και είμαι από τη Σικελία. Αν και έχω ζήσει στην Αυστραλία στο παρελθόν. Ε, τυχαία βρέθηκα εδώ, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι είμαι μονίμως σε επαφή με το πρόβλημα της ανεργίας. Βλέπω την ανεργία των νέων στη Σικελία καθημερινά. Και για εκείνους η Ευρώπη απέχει τόσο πολύ. Είναι τόσο μακριά. Πήγαινε στο σχολείο, παίρνουν διπλώματα, πτυχία, μάστερς πτυχιακά, κάνουν ό,τι μπορούν. Αλλά ε, δεν είναι σχεδόν άγνωστη η έννοια της εργασίας ε, ε, στους νέους αυτούς και δεν είναι μικρό το ποσοστό. Βλέπουμε καθημερινά τι τραβάνε για να βρουν δουλειά. Και μπορώ να σας πω ότι 80, ίσως και 90% των νέων μας στη δική μας περιφέρεια δεν έχει δουλειά. Χαίρομαι πολύ πραγματικά που βρίσκομαι εδώ σήμερα γιατί νομίζω ότι αυτές οι ανοιχτές ημέρες, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, θα πρέπει να έρθουν πιο κοντά στις περιφέρειες τους πολίτες που είναι τόσο μακριά. Και η Συγγελία είναι μία από αυτές τις περιφέρειες που απέχει τόσο πολύ. Εξεπλάγει σήμερα όταν είδα κάποιους Ιταλούς πολιτικούς που βγαίνουν συνέχεια στην τηλεόραση και λένε τι πρέπει να γίνει στην Ιταλία και ενώ σήμερα είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν εδώ σηκώθηκαν και έφυγαν. Εγώ είμαι τελείως ασήμαντη. Δεν είμαι κανένας, αλλά γνωρίζω τι συμβαίνει στα περισσότερα μέρη της Ιταλίας και η Σικελία όπου την χάνει να ζω και είμαι από τη Μεσίνη συγκεκριμένα. ναι, μπορεί να μένει στη Σικελία, αλλά έχετε δύο λεπτά μόνο για να μιλήσετε. Ε, ε, από τη Μεσίνη λέω, έρχομαι και σας παρακαλώ να κάνετε συγκεκριμένα πράγματα στην πράξη τα λόγια σας. Δεν βοηθούν τα λόγια τους νέους ούτε κανέναν άλλον πολίτη. Time for one more. έχει μείνει χρόνο για ένα μόνο τελευταίο μιλητή. Να σηκώσει παρακαλώ ψηλά το χέρι για να φανεί από το Προεδρείο. Τελευταία παρατήρηση ο κύριο 252. Λέγομαι Γιάννη Νέντελσον. Από τη Σουηδία. Εγώ ήμουνα δήμαρχο, μέλο ε, της Επιτροπής των Περιφερειών. Er. Ήμουν 11 χρόνια στην Επιτροπή των Περιφερειών, συμμετείχα στις ανοιχτές ημέρες. Ε, είναι εξαιρετική ευκαιρία διαλόγου, επιχειρηματολογίας, αλλά ακούγοντας τον Μισελ Ντελαμπάρ, να συμφωνήσω κι εγώ, δηλαδή διακομματικά, υπερκομματικά συμφωνούμε. Ε, το ίδιο και στην Επιτροπή της περιφερειακή ανάπτυξη. Συμφωνούμε με τον Επίτροπο, αλλά άλλοι επηρεάζουν την πολιτική και εκείνου πρέπει να πείσουμε. Πριν από 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τις περιφέρειες ε, για να γίνει διάλογος για την πολιτική συνοχή. Αλλά οι κυβερνήσει Και α πάρουμε τη Σουηδική κυβέρνηση για παράδειγμα. Δεν εισήλθαν σε διάλογο για το ίδιο ζήτημα με τι ε, περιφέρειε. Ακόμη περιμένουμε στη Σουηδία το διάλογο σχετικά με το πώ, πώς θα συμβάλλει αυτή η χώρα στην ε, περάτωση τη στρατηγική 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να το σκεφτεί αυτό σοβαρά. Οι κυβερνήσει είναι που πρέπει να ενεργοποιούνται στο διάλογο και να γίνει το διάλογο με τι περιφέρειε σε κάθε χώρα. Πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί αυστηρότεροι με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ντανούτα, πριν σου ξαναδώσω το λόγο, θα μπορούσα να δώσω το λόγο στην κυρία Μπρέσο και στον ε, Επίτροπο Χάν για να μας σχολιάσουν αυτά που ακούσαμε το απόγευμα. Κύριε Επίτροπε, θα θέλετε πρώτα εσείς μια σύντομη απάντηση. Ευχαριστώ. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, αυτές οι μέρες είτε τις λέτε open days, get together, connecting, ε, πρόκειται για ανταλλαγή εμπειριών, συναντήσεις. Αν θέλετε έρχεστε να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Αλλά μπορείτε και στον τομέα του ο καθένας να διοργανώσετε κάτι αντίστοιχο. Δεν σας εμποδίζει κανείς. Ε, το αντίθετο μάλιστα είναι ένα κίνητρο, ένα ένευσμα να γίνει αυτό. 260 ε, διοργανώσεις γίνονται. Είναι και ένα στοιχείο ε, που να λέμε όχι να τα κάνουν όλα οι Βρυξέλλες, από κοινού. Ο καθένας όπου του αναλογεί. Ο καθένας όπου έχει ευθύνες αναλάβει. Ακριβώς αυτή είναι δική μου έκκληση που θέλω να απευθύνω σε εσά. Και το δεύτερο, άκουσα τα όσα είπε ο Μισελ και οι άλλοι. Συμφωνούμε όλοι εδώ, αλλά γνωρίζουμε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν είναι και τόσο πεπισμένοι για το δίκαιο που έχουμε. Και εκεί θα πρέπει να δράσουμε και πολύ συχνά αυτή είναι υπεύθυνη ε, στις εθνικές κυβερνήσεις. Και εδώ θα πρέπει να δράσουμε ε, από τη μια η τοπική αυτοδιοίκηση και περιφερειακή και από άλλη οι Βρυξέλλες, να τους περικυκλώσουμε αν θέλετε και να πιέσουμε τις κυβερνήσεις. Ας αποκομίσουμε λοιπόν εμπειρίες, ε, ας ανταλλάξουμε απόψεις αυτές τις μέρες και να γυρίσουμε πιο ενισχυμένοι ε, στους τόπους μας για να αγωνιστούμε για την ευρωπαϊκή πολιτική και να τη διατηρήσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική στην περιφέρεια. Ε, Κυρία Μπρέσο. Καταρχάς, είναι γεγονός ότι σήμερα από ό,τι φαίνεται συμφωνούμε όλοι. Θυμάμαι όταν άρχισε η συζήτηση για την πολιτική συνοχή. Ήταν πολλές οι αμφιβολίες για τη σκοπιμότητα να διατηρηθεί ο στόχος της ανταγωνιστικότητας. Σήμερα σε ευρωπαϊκό ε, επίπεδο αυτός ο κίνδυνος φαίνεται να έχει αποσοβηθεί. Και ε, Νομίζω ότι είναι ήδη ένα αποτέλεσμα ε, των ε, ανοιχτών ημερών. Θα πρέπει να εδραιώσουμε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν έχει τελειώσει η συζήτηση για τη συνοχή ακόμα. Δεύτερη παρατήρηση. Ε, οι ανοιχτές ημέρες είναι βέβαια ένα βήμα διαλόγου. Μπορεί να γίνει στις Βρυξέλλες αλλά ε, γίνεται λόγος και ε, για τα πεπραγμένα, για τα όσα κάνουμε και θα κάνουμε στο μέλλον. Και στόχος είναι και σημαντικός ε, να βελτιώσουμε την εμπειρία μας και τη γνώση μας γυρνώντας πίσω τι έχουμε κάνει ο καθένα για να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών. Και είναι γεγονό ότι 6.000 παρόντες ε, είναι τοπικοί φορείς. Είναι φορεί από την τοπική αυτοδιοίκηση, εταίροι τη κοινωνίας των πολιτών και διαχειρίζονται την πολιτική συνοχή που όπως γνωρίζετε γίνεται σε εταιρικό ε, επίπεδο συνεργασία δηλαδή των οικονομικών και κοινωνικών δυνάμεων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ε, παρατήρηση τρίτη και για να έχουν μεγαλύτερη απήχηση αυτές οι μέρες, όχι μόνο εδώ στις Βρυξέλλες, αλλά να επεκταθεί και βέλειά τους να είναι παντού, καλούμε ε, όλους σας να διαδώσετε τα όσα θα πούμε εδώ και είπαμε ότι είναι 260 οι συνεδριάσεις που προβλέπονται, που έγιναν και θα γίνουν και συνδέονται με τις Open Days επιτόπου στις περιφέρειες προφανώς πάντα για να προβάλλουμε τα όσα έχουν γίνει και να συζητήσουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Δηλαδή δεν συζητούμε απλώς, ε, ε, διηγούμαστε τι έχουμε κάνει και ε, λέμε τι προτίθεται ο καθένας να κάνει. Ο καθένα στην περιφέρειά του και στην πόλη του. Και αυτό θα πρέπει να τα διαδίδουμε για να καταλαβαίνουν οι πολίτε ότι συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι χρήμα που έρχεται από το πουθενά, ε, αλλά είναι συνυπεύθυνη η Ευρώπη, μεγάλα έργα στην Ευρώπη και βλέπουμε τη δυνατότητα που έχει η Ευρώπη να διατηρήσει τα έργα αυτά και τη χρηματοδότηση. Να μην τερματιστεί αυτή η προσπάθεια. Γιατί ξέρουμε τι γίνεται ε, στα έργα που κρατάνε μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν μπορούν να ολοκληρώνονται γιατί σταματάει η χρηματοδότηση κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτές είναι οι ε, ανοιχτέ ημέρε να εξηγήσουμε όλοι στην Ευρώπη τι κάνουμε ο καθένας στον τόπο του και Τούμπαλιν να εξηγήσουμε ε, στις πόλεις και στις περιφέρειες τι κάνει η Ευρώπη. Και παρακαλώ όλους εκείνους που δεν το έχουν πράξει ακόμα για το επόμενο έτος να δηλώσουν ε, συμμετοχή για να διοργανώσουν ε, μία εκδήλωση με την κοινωνία των πολιτών, με τις κοινωνικές και οικονομικές δυνάμεις επιτόπου και να εξηγήσει ο καθένας τι έκανε. Και τελειώνω για τη Σικελία. Δεν μπαίνω στην ουσία του θέματος, αλλά ενθυμούμε ότι έχουν δικαίωμα οι πολίτες να ζητήσουν από του υπευθύνου να λογοδοτούν. Στη Σικελία πηγαίνουν πολλά ευρωπαϊκά χρήματα και θα πρέπει οι αρχές να λογοδοτούν στους πολίτες. Ευχαριστώ. Είμαι αμφιτρίων της ε, εναρκτήριας συνόδου, οπότε έχω και το πλεονέκτημα να κάνω τις καταληκτικές παρατηρήσεις. Ε, όπως ε, είπατε, μόλις αρχίσει η συζήτηση, θα επακολουθήσουν τρεις ημέρες ε, και είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε χρόνο για να ανταλλάξουμε εμπειρίες, παρατηρήσεις, ιδέες, που ζυμώνονται και πετάγονται σαν, σαν μανιτάρια σε αυτή την αίθουσα. Ε, θα είναι κέρια σημασία για το μέλλον τη περιφερειακή πολιτική, κέρια σημασία για όλε τι περιοχέ Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε να έχουμε οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή μέσω των καινοτομιών, των γνώσεων και τη καινοτομία, με τη ε, χρηστή διαχείριση των πόρων, τη ανάπτυξη που θα δημιουργήσουν τι νέε θέσει απασχόληση που προανέφεραν όλοι αυτό είναι ο βασικό μα στόχο και επίση να γίνει πιο ανταγωνιστική η Ευρώπη. Συμφωνήσαμε επίση ότι η συνθήκη προβλέπει ε, το στόχο αυτό τη πολιτική και αυτό εξακολουθεί να ισχύει, αλλά έχει σημειωθεί και μια αλλαγή την οποία οπωσδήποτε πρέπει να λάβουμε υπόψη. Οι περιφέρειες και οι πόλεις θα πρέπει να αντεπεξέλθουν όχι μόνο στι προκλήσει τη εσωτερική αγορά για τη ζώνη ενιαίου νομίσματος, αλλά θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν και στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, στον παγκόσμιο ανταγωνισμό ε, με τη μελλοντική οικονομική αρχιτεκτονική λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την εδαφική προγραμματικότητα μετά την ε, οικονομική κρίση σε περιφερειακό επίπεδο. Είναι απαραίτητο αυτό ούτως ώστε ε, να ε, μετικήσουν κάποιες περιοχές από την περίοδο υστέρηση στο μεταβατικό στάδιο και κατόπιν στο αναπτυξιακό στάδιο, τόσο ώστε να μεταβούν στο στόχο 2. Έτσι θα υποστηριχθούν οι προσπάθειες των ε, περιφερειών και νομίζω ότι θα πρέπει να παραμείνουν αναλύωτοι και στόχοι ως προς τη σύγκληση. Εδαφική συνοχή, ένα άλλο θέμα, ε, αναφέρθηκε μόνο επιγραμματικά ως ένα στόχος προς υλοποίηση, αλλά είναι ένα μέσο για να έχουμε καλύτερη ε, ανάπτυξη και ε, θα δώσει απαντήσεις σε όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει τώρα η Ευρώπη γιατί όλα έχουν μια εδαφική συνοχή και γι' αυτό η αξιολόγηση αντικτύπου για ε, την εδαφική πολιτική πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη λόγω και των ιδιαιτεροτήτων όλων των περιεχών Επίσης ε, το θέμα της αστικής ανάπτυξης ε, θα πρέπει να το δούμε από κοινού με όλες οι υπόλοιπες προκλήσεις. Τοπικές πρωτο... αναπτυξιακές πρωτοβουλίες όπως αυτές που ακούσαμε θα πρέπει να τονωθούν και οπωσδήποτε να ενισχυθεί η εδαφική και χωροταξική συνεργασία. Είπε κάποιος ότι πρέπει να άρουμε τους φραγμούς. λοιπόν με την εδαφική συνεργασία είναι ένα τρόπο, Είμαι πεπισμένη επίση ότι οι προτινόμε μεταρρυθμίσει τη πολιτική συνοχή θα μα οδηγήσουν στο μέλλον και θα μα οδηγήσουν σε μια πολιτική που θα στοχεύει σε απτά αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε φορά που το συζητάμε αυτό το θέμα το αναφέρει. Έτσι θα μπορέσουμε σε όλα τα επίπεδα τη διακυβέρνηση να δραστηριοποιηθούμε και νομίζω ότι η πολιτική θα πρέπει να βασίζεται με, σε μια επενδυτική στρατηγική προσανατολισμένη προς το μέλλον και τα απλά αποτελέσματα. Επίσης μην ξεχνάτε ότι έχουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για όλα τα διαρθρωτικά ταμεία και ο στόχος δεν είναι για να αποφύγουμε μόνο τις επικαλύψεις αλλά κυρίως για να χρησιμοποιήσουμε τις συνέργειες, να βασιστούμε σε κίνητρα στην αιρεσιμότητα, ε, στις, να προσανατολιστούμε προς τις πλέον αποτελεσματικές παρεμβάσεις ε, ε, η Ευρώπη 2020 συνιστά μεγάλη πρόκληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις εδαφικές ιδιαιτερότητες των επιμέρους περιεχών. Η Ευρώπη για να εκπληρώσει τους στόχους της, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να οδεύσει όλο ένα και περισσότερο προς νέους τρόπους χρηματοδότησης των επενδύσεών της. Έχει συσσωρευτεί εμπειρία αυτό, εμπειρία σε αυτό το τομέα και ο Φίλιπ Μέισταντ μας έδωσε απτά παραδείγματα, αλλά θα χρειαστούν και άλλες προσπάθειες, ε, ούτως ώστε να έχουμε μεγαλύτερη μόχλευση για τις δημόσιες επενδύσεις, κάτι που θα χρειαστούμε όλο ένα και περισσότερο στο μέλλον. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό. Θα πρέπει να γίνουν τα βασικότερα βήματα προ έναν πιο απλό αποτελεσματικό μηχανισμό. Με τη μεταρρύθμιση του 2006 και με την απλούστευση που επήλθε το 2008 και 2009, ανοίξαμε το δρόμο προς μια ευκολότερη, απλούστερη πολιτική, αλλά αυτή τη φορά θα πρέπει να είμαστε και πιο θαραλέοι για την απλούστευση. Αγαπητοί συναδελφοί, ε, Όπω είπε και η κυρία Φλολούκα, ε, να κάνω και εγώ ένα σχετικό σχόλιο. Στο, στο κτίριο Σαγλεμάνια πριν από πέντε χρόνια είχαν έρθει χιλιάδε άνθρωποι από τι ε, περιφέρειε τη Ευρώπη και αποφασίσαμε την ε, στρατηγική τη Λισαβόνα να την κατεβάσουμε σε εισαγωγικά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Και τότε είχατε πει ότι η περιφερειακή πολιτική οδήγησε στο να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια σε σχέση με τη στρατηγική τη Λισαβόνα Λισαβόνας και με τη σημερινή ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, μπορούμε να πούμε ότι η μοναδική επιτυχή σε διάσταση της στρατηγικής Λισαβόνας ήταν η περιφερειακή πολιτική. Λοιπόν, ας χρησιμοποιήσουμε την στρατηγική Ευρώπη 2020 και κυρίως αυτές τις βασικές πρωτοβουλίες επωνομαζόμενες flagship initiatives να τις ε, τοποθετήσουμε σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και σίγουρα ε, θα ε, τελεσφορήσουν οι προσπάθειές μας. Τα εδαφικά σύμφωνα, τα τοπικά σύμφωνα, τα προαναφέρατε, θα είναι εξαιρετική κοινωνική πλατφόρμα ώστε η Ευρώπη 2020 να βοηθήσει την Ευρώπη. Κλείνοντα, ε, θα έλεγα ότι επιτέλου θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το να διευρύνουμε την Ευρώπη πέρα από το ευρωπαϊκό επίπεδο διακυβέρνηση, εμπλέκοντα τι τοπικέ αρχέ, εμπλέκοντα τι περιφέρειε, τι πόλει, τα χωριά, αυτό έχει ω αποτέλεσμα όχι μόνο να έρχονται πιο κοντά οι πολίτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά διευρύνει και την ίδια, μεγενθύνει αν θέλετε την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να είναι χρήσιμη η εβδομάδα που θα ακολουθήσει και όπως είπε ο κύριος Μισελ Ντελμπάρ έχουμε πολλά να κάνουμε και εκτός της αιθούσης ε, σε όλα τα όργανα, σε όλα τα πλαίσια στα οποία λειτουργούμε πρέπει να εξηγούμε σε αυτούς που δεν γνωρίζουν αλλά και σε αυτούς που γνωρίζουν την περιφερειακή πολιτική, γνωρίζουν τα αποτελέσματά τους αλλά δεν καταλαβαίνουν ή δεν θέλουν να καταλάβουν. Ας τους μιλήσουμε λοιπόν ούτως ώστε η πολιτική συνοχή μετά το 2013 ε, να ε, λειτουργήσει πλήρως προς όφελος των πολιτών και να βελτιώσει την Ευρώπη. Με αυτά τα λόγια θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την υπομονή που μείνατε εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ τους ε, ε σύνοικοδεσπότες μου. Σας ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Βρήκατε όλοι χρόνο για να έρθετε να μιλήσετε. Δεν είχαμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Τα καταφέραμε. Καλή εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Ελία τη συνεδρίαση.